Καλώς ορίσατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ζητώ συγγνώμη για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση. Χρειαστήκαμε λίγο περισσότερο χρόνο με τους συντονιστές. Σας καλωσορίζω και ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις μας σήμερα το πρωί. Το πρώτο σημείο Φέρει επί των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης την ισότητα των φύλων. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Καλωσορίζω την κυρία Όσνατ Λουμπράνη. Είναι η διευθύντρια του Αναπτυξιακού Ταμείου του ΟΗΕ για τις γυναίκες ε, UNIFEM χρησιμοποιείται το ακρόνιμο αυτό. Σας ε, καλωσορίζουμε. Ε, θα σας δώσουμε το λόγο για την παρουσίασή σας περίπου ε, ένα τεταρτάκι και στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση. Θα υποβληθούν οι ερωτήσεις από τα μέλη και το καθεξής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Είναι μεγάλο προνόμιο για μένα και για τη UNIFEM να είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών που μου δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστούμε μαζί σας κάποια στοιχεία, τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει για την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις ε, επιπτώσεις για την ε, θέματα ισότητας των φύλων. Οι πληροφορίες ε, είναι από διάφορα στοιχεία. Με χαρά αργότερα να σας δώσω τον πλήρη κατάλογο των ε, αναφορών. Αλλά να σας πω καταρχάς ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα δεδομένα για τα αποτελέσματα της κρίσης. Κάποια από τα στοιχεία της ανάλυσης ε, είναι από αναλύσεις που έχουμε από προηγούμενες κρίσεις, δεδομένα δηλαδή τα οποία έχουμε συλλέξει από εκεί. Να σας πω λοιπόν ότι η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι 50 εκατομμύρια άτομα μπορεί να απληχθούν από τη ε, φτώχεια ε, λόγω της ύφεση ε, με ένα εκατομμύριο ακόμα τα οποία φτάνουν στη φτώχεια το 2008. εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάνουν το εισόδημό τους, τις δουλειές τους και παλεύουν για να επιβιώσουν. Από ό,τι ακούσαμε και χθε τι ειδήσει, άκουγα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και κάποιε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουν ε, να λένε ότι ξεκινάει η ανάκαμψη, που είναι καλό νέο, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζεται και το γεγονό ότι δεν έχουμε ξεφύγει από το σκόπελο ακόμα και ότι η ανάκτηση κατά πάσα πιθανότητα δεν θα φτάσει στου ανθρώπου που έχουν πληχθεί περισσότερο. όχι μόνο για την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε και σε αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν λιγότερες ικανότητες να εφαρμόσουν μέσα αντα, ε, ανταπόκριση στην κρίση. Το θέμα των ε, στόχων της χιλιετίας είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν φαίνεται να προχωρούν και σήμερα εγώ θα σας πω πώς επηρεάζει τις γυναίκες και τα κορίτσια το θέμα αυτό. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία ως προς την ε, διαθέσιμη ε, παροχή υγείας, ε, κυρίως ποιοτική και επίσης μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα τα οποία μπορεί να περιορίσουν ακόμα τις περισσότερο τις δυνατότητές τους για πληρωμένη εργασία. Επίσης, η... τα κορίτσια κατά πάσα πιθανότητα στις φτωχές χώρες μπορεί να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν το σχολείο γιατί οι φτωχότερες οικογένειες ε, δεν έχουν αρκετούς πόρους για να τη στείλουν σχολείο. Το 2000 τα κορίτσια ήταν το 54% του πληθυσμού που εγκατέλειπε στο σχολείο. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το ποσοστό θα ανέβει και μπορεί ε, περισσότερα από αυτά τα κορίτσια να μην επιστρέψουν ποτέ στο σχολείο. Είναι προφανές λοιπόν ότι ένας τομέας ο οποίος ε, θα αλλάξει ριζικά ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης είναι η απασχόληση. Θα διαπιστώσουμε ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες ε, βγάζουν τα προστοζήν τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες υπάρχει πιθανότητα να χρειαστούν χρόνια για να ανακάμψει ο χώρος της απασχόλησης και σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην παρέχει την οικονομική ασφάλεια η οποία είναι απαραίτητη για την ευζοία τους. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες κρίσεις όπου οι οικονομίες ανέκαμψαν πολύ γρήγορα, αυτή τη φορά ουσιαστικά καταραίει η παγκόσμια ζήτηση και πολλές βιομηχανίες δυσκολεύονται να επιζήσουν και γενικότερα ε, το περιβάλλον θα αλλάξει άρδινε στον τομέα αυτό και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις χώρες τόσο ώστε να ξαναρχίσουν να δουλεύουν οι άνθρωποι και... σε διάφορες ε, θέσεις και να μπορέσουν να επανακτήσουν τις θέσεις εργασίας. Η έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, λέγει ότι περίπου 40% των εργαζομένων διεθνώς είναι γυναίκες. Στην αρχή οι άντρες ε, οι άντρες ε, ε, είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας αλλά βλέπουμε τώρα ότι ενώ αρχίζει να επιβραδύνεται ο ρυθμός της ε, απολύας θέσεων εργασίας στους άντρες αυξάνεται στις γυναίκες και έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό για τις γυναίκες τώρα από ό,τι για τους άντρες αυτό βέβαια θέτει σε κίνδυνο τα κεκτημένα όσον αφορά την ισότητα των ε, φύλων τόσο ε, και στις οικογένειες όσο και στις θέσεις εργασίας. Υπάρχουν ε, βιομηχανίες όπου οι γυναίκες είναι 70-80% των εργαζομένων και σήμερα έχει ε, αποδεκατιστεί το ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποιείται ιδίως ε, στον τομέα παραδείγματος χάρη των ηλεκτρονικών διότι ίσως ε, θυμάστε την περίπτωση που αναφέρθηκε στην Νοτιοανατολική Ασία αλλά και στη Νότιο Αφρική υπήρχαν ε, ε, επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούσαν πολλές γυναίκες από το 2002 αλλά τώρα έκλεισαν στο Λεσότο και σε άλλες χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι γυναίκες επίσης ήταν το 85% των απολυμένων εργαζομένων και στην Ανατολική Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχει μία παρεμφερής ε, κατάσταση ε, δηλαδή έχουμε 40.000 άτομα τα οποία απολύθηκαν στον ε, τομέα της κλωστοϊφαντουργίας και των ενδυμάτων εκ των οποίων το 90% ήταν ε, γυναίκες και αυτό οφείλεται εις ε, ε, την οικονομική κρίση. Το ίμιση των εργαζομένων σήμερα διεθνώς εργάζεται χωρίς επίσημο συμβόλαιο εργασίας και αυτό το ποσοστό θα, ε, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Εδώ πρόκειται για μια έκθεση του ΟΣΑ όπου λέγεται ότι οι περισσότερες γυναίκες ε, οι οποίες εργάζονται σε ε, θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας θα πληγούν περισσότερο όπως παραδείγματος χάρη οι μετανάστες εργαζόμενοι ε, που κινούνται από την ε, Αφρική προς την Νότιο Αμερική. Ε, υπάρχουν γενικώ διάφορες τάσεις μετανάστευσης και πολλοί αναγκάζονται να γυρίσουν στις χώρες τους γιατί δεν μπορούν να στέλνουν ε, χρήματα. Στις χώρες της Κεντρικής Ασίας έχουν μειωθεί σημαντικά οι θέσεις εργασίας ε, σε σχέση με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Στις ε, χώρες προορισμού στην Αμερική επίσης υπάρχει μία αύξηση μετανάστευσης διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ψάχνουν ακόμη δουλειά εκτός της χώρας τους αλλά ενδέχεται να αλλάξει αυτή η τάση διότι κλείνουν τα σύνορα για τους μετανάστες σε πολλά κράτη όπως παραδείγματος χάρη ή στην Ισπανία κατόπιν της στον τουρισμό πολυτελείας και ε, ιδίως ε, για τις γυναίκες που προερχόντουσαν από την Λατινική Αμερική και είχαν μεταναστεύσει. Υπάρχει λοιπόν μία παραοικονομία η οποία προσπαθεί να επιβιώσει και εκεί ακόμη οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο διότι ε, έχουν άτακτα ωράρια και ανεπαρκή πληρωμή. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω ε, λίγο και να σχολιάσω τη διασύνδεση μεταξύ οικονομικής ε, ε, κρίσεως και βίας υπάρχει δηλαδή μία διασύνδεση μεταξύ της ε, οικονομικής αστάθειας και της βίας κατά των γυναικών. Υπάρχει ένα έγγραφο σχετικά με αυτά ε, τα θέματα ε, της, βίας κατά των γυναικών και με στην οικογένεια και σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ε, ανοιχτές γραμμές ε, γιατί διαπιστώνεται και πάλι μία τέτοια τάση και διαπιστώνουμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες αυξάνονται πολύ οι γυναίκες οι οποίες ζητούν βοήθεια και αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο με την ε, έλευση της κρίσεως. Ε, η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ε, αναφέρει στην έκθεσή της ε, τις περιπτώσεις βίας ε, των, κατά των γυναικών και ότι αυτές είναι συνδεδεμένες με την οικονομική κρίση. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ και βλέπουμε ότι ε, όταν υπάρχουν μειώσεις ή μειώσεις ε, στην αμοιβή πλήττουν πρώτα τις ε, κοπέλες και μετά τους άνδρες η υγεία επίσης των γυναικών και των νέων κοριτσιών κινδυνεύει πολύ περισσότερο τώρα διότι όλο περισσότερες γυναίκες ε, δεν ε, συμβουλεύονται πλέον ε, ιδιωτικά ένα γιατρό αλλά βασίζονται στη δημόσια υγεία η οποία βρίσκεται σε κατάρρευση και είναι υπερβολικά επιβαρημένη. Έχουμε λοιπόν προβλήματα όχι μόνο στην Αφρική αλλά και στην Κεντρική Ασία και ακόμη και στην Ευρώπη ο τρόπος με τον οποίο ε, ε, επηρεάζει η κρίση τις γυναίκες είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να το εξετάσουμε διότι στην Ασία και στον Ειρηνικό έχουν προβλεφθεί δύο μέτρα καταρχήν ε, αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δεύτερον ε, προστασία ε, των γυναικών και των οικογενειών από την κρίση και εφόσον οι περισσότερες δημόσιες επενδύσεις αναφέρονται στις διαρθρωτικές δαπάνες υποδομής πρέπει να δούμε ε, πώς ε, ε, κατανέμονται αυτές οι δαπάνες και στις, στα έργα υποδομών συνήθως τις εργασίες αυτές τις αναλαμβάνουν άνδρες και οι γυναίκες αναλαμβάνουν μόνο δευτερεύουσες θέσεις. Ε, επίσης εξετάσαμε την χρηματοδότηση σχολείων, νοσοκομείων και άλλων οργανισμών που μπορεί να είναι προς όφελος επίσης ε, των ε, γυναικών. Εξετάσαμε επίσης τους βρεφικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία όπου οι γυναίκες είναι χρήσιμες. Ε, πρέπει να δούμε επίσης ποιος θα υποφεληθεί αν ο δρόμος που κατασκευάζεται θα βοηθήσει τις γυναίκες να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά και τα παιδιά στα σχολεία. Ε, θα υπάρχει χρηματοδότηση για να επανδρωθούν ε, τα ιδρύματα αυτά, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και πρέπει να δούμε και ποιες βιομηχανίες πρόκειται να βοηθηθούν διότι έχουμε ακούσει ότι ε, βοηθούν τις τράπεζες αλλά το ερώτημα είναι τα χρήματα απευθύνονται στις βιομηχανίες. Ποιες βιομηχανίες χρησιμοποιούμε διότι έχουμε ακούσει για την αυτοκινητοβιομηχανία σε διάφορες χώρες αλλά έχουμε κοιτάξει και άλλα παραδείγματα όπου ε, οι βιομηχανίες στο Βιετνάμ και στην Ταϊλάνδη ε, αποβλέπουν εις ε, την στήριξη ε, μικρών επιχειρήσεων ε, αντί για ε, τις χειροτεχνικές επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι οι θέσεις ε, των γυναικών μειώνονται αλλά έπρεπε επίσης να δούμε εάν υπάρχουν φορολογικές απαραλλαγές εάν υπάρχει χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις για γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα σε διάφορες χώρες διότι στην Αργεντινή παραδείγματος χάρη ε, υπάρχει προσπάθεια να ενταχθούν οι γυναίκες στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων και αυτή η πολιτική είναι υπέρ των γυναικών. Θα έπρεπε επίσης να πούμε ότι πρέπει να δούμε τι πόροι απευθύνονται σε κάθε κατηγορία διότι συζητήσαμε με διάφορα υπουργεία για να ε, μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα υποφεληθούν εξίσου με τους άνδρες και όσον αφορά την ε, παρακολούθηση θα πρέπει ε, να δούμε μέχρι ποιου σημείου η, η, τράπεζα η Διεθνή Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενδιαφέρονται να στηρίξουν τις γυναίκες στις υποανάπτυξη χώρες πώς βοηθούνται αυτές διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ προσπαθούν να καταρτήσουν ένα πρόγραμμα κατά τρόπον ώστε όλοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις να υπάρχει άμεση χρηματοδότηση εις ε, τις ε, αγρότησες να υπάρξουν ε, χρηματοδοτήσεις ε, για τις ε, μικρές αγροτικές επιχειρήσεις τις οποίες διαχειρίζονται γυναίκες, να υπάρξει αύξηση εργασίας στον τομέα της περίθαλψης και της παιδείας και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας χωρίς εκμεταλλεύσεις σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός γυναικών. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας μόνο για τους άντρες και κοινωνικά επιδόματα μόνο για τις γυναίκες Υπάρχει μία άτακτη διεθνής αγορά η οποία δίνει την ευκαιρία συγχρόνως να υπάρξει αλλαγή και είναι αλλαγή την οποία πρέπει να υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις διότι ε, ε, μία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας λέγει ότι ε, ε, τα ωφέλη από την δημιουργία θέσεων εργασίας για γυναίκες μπορεί να έχει μακροοικονομικά πολύ καλά αποτελέσματα και θα μπορέσουν να προλάβουν την μελλοντική φτώχεια γι' αυτό και θα πρέπει τα μέτρα αυτά να ληφθούν γρήγορα. Επειδή όμως αναμένεται ότι οι επιπτώσεις στην απασχόληση θα είναι πιο σημαντικές, θα πρέπει όλοι να ξανασκεφθούν ορισμένες οικονομικές ε, ιδέες οι οποίες ε, είχαν αποκρισταλωθεί στα οικονομικά πρότυπα του 19ου και 20ου αιώνα. Δηλαδή ε, θα πρέπει η οικονομική παραγωγή να ανταποκριθεί στις κλιματολογικές αλλαγές. Θα πρέπει να προωθήσουμε την πράσινη οικονομία η οποία θα μπορέσει να είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη στο μέλλον και τα κίνητρα που θα διατυπωθούν δεν θα πρέπει να βασίζονται στη φθηνή εργασία των γυναικών. Θα πρέπει οι γυναίκες να είναι εκπαιδευμένες για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με τους άντρες και όσο οι υποανάπτυξη χώρες αναπτύσσουν την γεωργία και την οικονομία της υπαίθρου θα μπορέσουν να προβούν σε μία επανάσταση βασισμένη στις γυναίκες οι οποίες θα πάψουν να εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και την εξάρτησή τους από τις διεθνείς αγορές. Ε, για να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι υπόλογες οι κυβερνήσεις και η τελευταία έκθεση η οποία έχει καταρτιστεί διεθνώς επ' αυτού ε, αποδεικνύει ότι ε, ο δημόσιος ε, τομέας ε, δεν είναι υπόλογος σε κανένα σε σε πάρα πολλές χώρες και γι' αυτό αυτό ισχύει από τις τράπεζες μέχρι ε, διάφορους οργανισμούς και τέλος το διεθνές οικονομικό σύστημα. Δεν είναι απαραίτητο να ισχύσει αυτό διότι ζητούμε από τις χώρες να μπορέσουν να αναδιατυπώσουν το σύστημα το οποίο μπορεί να προωθήσει την ισότητα των φύλων και μέτρα τα οποία θα περιλαμβάνουν υπεύθυνο προϋπολογισμό και καλύτερα κέντρα περιθάλψεως παιδιών που θα χρηματοδοτούνται από το δημόσιο κατά τρόπον ώστε οι γυναίκες να μην χρειάζονται εξωτερική βοήθεια και να μπορέσουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Και ολοκληρώνω γι' αυτό σε τέτοιες εποχές κατέρευσαν τα πρότυπα και είναι δύσκολο να υπάρξει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ένα προβλέψιμο μέλλον και τελειώνω εδώ και σας ευχαριστώ. Ehm, σας ευχαριστούμε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής, σχόλια και παρατηρήσεις. Θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε και να σχολιάσετε τις παρεμβάσεις των μελών. Η κυρία Γκιουμάγια, στη συνέχεια εγώ, η κυρία Τόμσον. Η κυρία Γκιουμάγια θα πάρει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω στην έδρα, διότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία ως αντιπρόεδροι με τη συναδέλφους από την προηγούμενη θητεία. Επομένως χαίρομαι που σας βλέπω, Πρόεδρο να καλωσορίσω τη Διευθύντρια. Ξέρω ότι έχει τεράστια πείρα στα θέματα αυτά και χαίρομαι που βλέπετε και πόσο επαγγελματικά συμπεριφέρεται. Νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε και πρέπει να φαινόμαστε επαγγελματίες. Δεν αρκεί βέβαια αυτό, πρέπει να είμαστε και επαγγελματίες. Τώρα, για την οικονομική κρίση. Ταξιδεύανα την Ευρώπη συζητώντας το θέμα και αρχίσαμε να συζητάμε τις γυναίκες και την κρίση την πρώτη φορά στο Παρίσι στις 19 Μαρτίου και εκεί διαπιστώσαμε ότι το 80% των ανδρών πλήττονται από την ε, κρίση. Και από εκεί κατέστη σαφές ότι επειδή δεν μπορούμε να τα ε, σκεφτούμε μακροπρόθεσμα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία, διότι όμα το σκεφτείτε μακροπρόθεσμα, η κρίση αυτή αφορά και τις γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν για την κρίση να δούμε τι γίνεται με θέματα ε, απασχόληση, τι γίνεται με το θέματα, την απουσία γυναικών σε κάποιου τομεί. Αν δείτε για παράδειγμα τον κατασκευαστικό τομέα, οι περισσότεροι είναι άνδρες. Τώρα, για το θέμα των τραπεζών θα πρέπει να υπάρχουν πολύ σαφείς δράσεις. Οι τράπεζες έχουν δικλείδες ασφαλείας, αλλά θα πρέπει να δουν και τι γίνεται αργότερα. Για τους πελάτες θα πρέπει να δίνονται διαφορετικά δάνεια, πιο μακροπρόθεσμα και να δούμε τι υπάρχουν. Διότι εξακολουθεί να υπάρχει, αν εξακολουθεί να υπάρχει κέρδος από τις τράπεζες και οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ε, αφήσουμε τις τράπεζες να το κάνουν αυτό. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα της εξωτερικής ανάθεσης. Ε, πάνω των 80% των θέσεων απασχόλησης στον τομέα αυτό είναι γυναίκες. Τώρα για τις φορολογικοαπαλλαγές και το δημόσιο τομέα ε, βλέπετε ότι αναμένεται και αύξηση της ανεργίας για τις γυναίκες. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε για τις ε, ε, γυναίκες και τις οικογένειές τους και το πώς βιώνουν αυτές την Κρήτη και αν τα δείτε από αυτή την οπτική θα διαπιστώσετε ότι και στη Νέα Υόρκη υπήρχε μία διάσκεψη που συζητήθηκε η κατάσταση των γυναικών. Ε, νομίζω ότι οι οικογένειες αυτές είναι διαφορετικές. Πρέπει να είμαστε ε, προετοιμασμένοι για τις νέες δομές οικογένειες διότι η κλασική οικογένεια δεν υπάρχει ε, πλέον και Το θέμα της άδεια μητρότητας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η κυρία Λουμπράνη αναφέρθηκε και για τις, στις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το χάσμα της ένδυας αυξάνεται και οι γυναίκες πλήττονται πάρα πολύ από την ένδυα. Οι περικοπές στον προϋπολογισμό είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και φιλανθρωπικό έργο και αλληλεγγύη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα για την κατάσταση των γυναικών ε, και την αντιμετώπιση της κρίσης. Πρέπει να επενδύσουμε στο δημόσιο τομέα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ε, και κοινωνικές δομές. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, το διαχωρισμό που γίνεται, διότι αν δείτε η κρίση είναι λιγότερη αποτελεσματική αν δεν υπάρχουν γυναίκες στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν δύο γυναίκες οι οποίες διευθύνουν τράπεζες και η κρίση στις τράπεζες αυτές δεν ήταν τόσο μεγάλη. Βλέπουμε ότι πρέπει να ε, προβλέπονται περικοπές στον προπολογισμό για τα θέματα ισότητας του φύλου και προπολογισμό για το φύλο. Επομένως δεν θα πρέπει να αφήσουμε να γίνει αυτό και όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς μας. Αυτές λοιπόν ήταν οι προτάσεις μου και οι ανησυχίες και πιστεύω στεναρά ότι πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού Χαίρομαι που γνωρίζω κάποιους από εσά, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω, αλλά αυτή τη στιγμή ε, είμαι σε διαφορετική θέση. Ε, είμαι πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και ελπίζω τα θέματα ισότητας των φίλων να τεθούν στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις απόψεις. Ε, θα ήθελα και εγώ να παρατηρήσω κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδοθούν οι ευθύνες για την οικονομική κρίση που γνωρίζει η κοινωνία μας. Όταν υπέρχεται μια τέτοια κρίση, ε, σημαίνει όμως επίσης ότι ε, μπορεί να σημειωθεί και κάποια αλλαγή. Είναι μια πρόκληση και μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή. Ε, στον τομέα της οικονομίας, ευελπιστούμε ότι θα σημειωθεί αλλαγή ε, σε σχέση με την εξουσία στην παγκόσμια οικονομία, στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ε, όπου ε, δεν είχε προβληθεί ε, μέχρι στιγμής επαρκώς η εικόνα και ο ρόλος των γυναικών ε, καθώς και το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Με τη σημερινή συζήτηση βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, δηλαδή με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε την κρίση, να την αναδείξουμε σε μια πρόκληση που θα μας οδηγήσει σε καλύτερη μελλοντική δράση διαπιστώνουμε τις ζημιές ε, της κρίσης, αλλά δεν θέλουμε να επανέλθει όπως γίνεται συνήθως η κατάσταση ε, στα προηγούμενα δεδομένα. Δεν θέλουμε να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για να επέλθει αλλαγή. Γιατί τον τομέα των υπηρεσιών, Τώρα, μιλήσαμε για το κατά πόσο ε, ε, επλήγησαν οι εξαγωγές λόγω της κρίσης και φαίνεται ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα σημειωθεί και μελλοντικά στον τομέα των ε, υπηρεσιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας για την απασχόληση των γυναικών θα μπορούσατε να σχολιάσετε τις επιπτώσεις της κρίσης επί του τομέα των υπηρεσιών. Η κυρία Τόμσεν και στη συνέχεια η κυρία Γιαβόκα. Η κυρία Τόμσον πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. για τα πακέτα επενδύσεων βλέπουμε ότι τα ε, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με αυτά τα πακέτα αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους άντρες στην Ευρώπη δεν συζητείται το θέμα των επιπτώσεων της κρίσης επί των γυναικών και επί των θέσεων εργασίας για τις γυναίκες. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο, αυτά που είπατε περί πράσινης οικονομίας. Εμείς ε, στο Κοινοβούλιο συζητάμε για την ε, ε, δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, στο τομέα του περιβάλλοντος και το φθινόπωρο η Σουηδική Προεδρία μας έκανε μια πρόταση για μια νέα οικο-οικονομία, πράσινη οικονομία, ε, πρόγραμμα που θα, ε, στο οποίο θα πάρει τη σκητάλη μετά η Ισπανική Προεδρία. Ε, υπάρχει σοβαρός διχασμός στην αγορά εργασίας ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες γιατί στον ενεργειακό τομέα σήμερα στην Ευρώπη το 80% είναι θέσεις εργασίας για τους άντρες. Και θέλω την άποψή σας επ' αυτού. Πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε αυτή την κρίση για να μην είναι τόσο διχασμένη η αγορά εργασίας, διχοτομημένη ανάμεσα στους άντρες και στις ε, γυναίκες. Σας ευχαριστώ κυρία Τόμσον, η κυρία Γιαρούκα και μετά η κυρία Παβανόβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ακούσαμε πάρα πολύ καλέ πληροφορίες, μπορέσαμε να διαπιστώσουμε πώς έχει κατάσταση. Αυτό που με ανησυχεί και αυτό που καταδεικνύεται περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι ότι οι οικογένειε που ούτω ή άλλω ήταν φτωχέ έχουν πληχθεί τόσο ανεπανέρθετα που τα περισσότερα παιδιά τους ε, βρίσκονται πλέον σε ιδρύματα και αυξάνεται συνέχεια ο αριθμό. Και αυτό φαίνεται ότι θα είναι το δυσκολότερο πρόβλημα. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οι οικογένειες αυτές είναι συνήθως μεγάλες οικογένειες. Πολύ συχνά οι μόνοι που εξοικονομούν τα προστοζούν στο σπίτι είναι οι γυναίκες, διότι στην μετακομμουνιστική ε, εποχή ε, οι άνδρες ε, ε, είχαν, συγκεκριμένε, είχαν ήδη χάσει τη δουλειά τους και οι μόνες που μπορούσαν να ε, κάνουν μαύρη άτυπη εργασία ήταν οι γυναίκες. Αυτές λοιπόν είναι οι γυναίκες οι οποίες χάνονται ουσιαστικά και το μεγαλύτερο πρόβλημα που διαπιστώνω είναι ότι στις οικογένειε οι οποίες υπάρχει έστω και ένας ο οποίο εξοικονομεί τα προστοζήν είναι αυτοί που χάνουν τη δουλειά τους. Ε, οι άστεγοι αυξάνονται και οι οικογένειες χάνουν τα σπίτια τους, όχι μόνο άτομα. Πώς θα ανταποκριθούν λοιπόν οι διάφορες χώρες αυτό, διότι από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή από τα προγράμματα ανάκτησης, μας ανησυχούν ε, οι απώλειες θέσει εργασίας από τη μεσαία τάξη, που είναι φυσικά ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά ρίχνουμε πάρα πολύ το βάρος αυτούς και ξεχνάμε τους ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, που πεινούν. Πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ουγγαρία περίπου 3 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται στην ε, γραμμή της ένδυας και 300 περίπου χιλιάδες άτομα ε, είναι από και είναι τα άτομα τα οποία κυρίως πεινούν. Μιλάμε για 800.000 ανθρώπους περίπου και δεν βλέπουμε και ιδέες από τις κυβερνήσεις για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα ευχαριστούμε κυρία Γιαρόκα. Η κυρία Παβανόβα τώρα. Ευχαριστώ. Uh, uh, Εντυπωσιάστηκα από την παρουσίασή σας. Είναι σαφές σε όλους ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης υπάρχουν διακρίσεις και οι γυναίκες χάνουν περισσότερες δουλειές. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση για τρεις πολύ συγκεκριμένες ε, ομάδες. Η μία, όπως είπε και η συνάδελφος, η κυρία Γιαρόκα, είναι οι γυναίκες από μειονότητες. Έχετε δεδομένα, έχετε στοιχεία τα οποία μπορεί να σας δίνουν μια καλύτερη εικόνα ε, από τις γυναίκες που απολύονται κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουμε περισσότερες γυναίκες στην, ε, ε στις μειονοτικές ομάδες ε, και οι γυναίκες με αναπηρία. Μπορούν να τεθούν επίσης όροι στην αγορά εργασίας. Υπάρχει μια διπλή διάκριση. Γυναίκες και ιδίω ε, γυναίκες με αναπηρία, περισσότερες γυναίκες με αναπηρία χάνουν τις δουλειές τους. Και τρίτον, η τρίτη ομάδα που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη είναι οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και σκοπεύουν να κάνουν παιδί ή γυναίκες οι οποίες ε, κάνουν θεραπείες ε, αναπαραγωγικής ε, υγείας. Πολλές γυναίκες ε, σε ηλικία τέτοια χάνουν τη δουλειά τους από τα στοιχεία που έχω και ένα 30% κρύβουν το γεγονός ότι έχουν πρόθεση να κάνουν παιδί. Έχετε στοιχεία γι' αυτό. Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε αυτές τις τρεις τόσο ευάλωτες ομάδες. Και μία πρόταση Ε, και ερώτηση και πρόταση. Υπάρχουν πρωτοβουλίε και υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν προγράμματα για να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα για τι γυναίκε. Και πώ μπορεί να γίνει αυτό, ξεκινώντα από την κατάλληλη παιδεία, επιμόρφωση, αύξηση τη πείρα του, για να μπορέσουν ε, ίσω να ε, είναι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας, κυρίως για ε, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, διότι φαίνεται ότι πλέον οι γυναίκες θεωρούνται καταλληλότερες για υπηρεσίες και όχι για επαγγέλματα υψηλού προφίλ, αλλά υπάρχουν ε, επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται στην κοροφή, κορυφή και είναι πολύ ανταγωνιστικά όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, πληροφορική, ε, χρηματοοικονομικά, συμβούλων. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να εντείνουμε και τις προσπάθειές μας για να ε, λάβουν οι γυναίκες θέσεις εργασία σε αυτά τα επαγγέλματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Παβανόβα, η κυρία Μπάουερ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να διευρύνω λίγο το πεδίο της συζήτησης. Είχαμε κάποια εμπειρία ε, και κάποιες αυξημένες γνώσεις σχετικά με την ε, αύξηση της βίας και της επιθετικότητας λόγω της κρίσης. Έχετε κάποια σχετικά δεδομένα, μήπως ε, έχετε δικές σας εμπειρίες σε αυτό το τομέα. Ε, είναι σοβαρές, ε, ε, μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρές οι παρενέργειες της κρίσης. Κάτι άλλο τώρα, υπάρχει κάποια πρωτοβουλία για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή απόκτηση αυξημένων οικονομικών γνώσεων. Ενίσχυση του οικονομικού κομματιού της διδακτικής ε, ύλης, δηλαδή, διότι λόγω της κρίσης διαπιστώσαμε ένα κενό γνώσεων ε, που υπάρχει. Έλλειψη γνώσεων σε σχέση με το τι συμβαίνει στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε σχέση με το πώς επηρεάζει μια τέτοια κρίση στην καθημερινή τους ζωή. Υπάρχει κάτι σχετικό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Η κυρία Μάισερ τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και κυρία Λουμπράνη σε εσάς για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η κυρία Παβάνοβα και ε, μπορείτε ίσως και εσείς ε, να το επιβεβαιώσετε ότι υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στις νέες τεχνολογίες και στις ε, υψηλές τεχνολογίες όπου δεν είναι υποχρεωτικά ότι οι θέσεις αυτές είναι θέσεις ανδρών, υπάρχουν και γυναίκες που μπορούν να τις καλύψουν και αυτό έχει σχέση με την παιδεία και με το ενδιαφέρον για τεχνικές, ε, ε, τεχνικά επαγγέλματα και τεχνολογίες. Υπάρχουν λοιπόν ε, προγράμματα όπου προσπαθεί κανείς στα σχολεία ήδη να ξυπνήσει την περιέργεια των κοριτσιών για τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία γιατί τα κορίτσια συνήθως ενδιαφέρονται για άλλα θέματα. Έχετε κάνει κανένα πρόγραμμα για να ξυπνήσετε αυτά τα ενδιαφέροντα γιατί πιστεύω πιστεύω ότι και οι γυναίκες ε, και τα κορίτσια μπορούν ε, να είναι εξίσου αποτελεσματικοί όπως και οι άντρες στους τεχνολογικούς τομείς. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σαμπόσκα είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Διευθύντρια για την περιστατωμένη και ενδιαφέρουσα έκθεση που μας παρουσίασε. Εσείς εκπροσωπείτε τον ΟΗΕ στην Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο, οπότε κανονικά θα παρακολουθείτε την ε, στήριξη που δίνετε στους πλέον ισχυρούς στην Ευρώπη Πιστεύετε ότι χρησιμοποιούνται ορθώς τα κονδύλια γιατί το μεγαλύτερο μέρος τους έχει ενισχύσει τους ήδη ισχυρούς και όχι τις ευτοχότερες χώρες. Επίσης, ε, κατά τη διάρκεια ε, της οικονομικής ε, κρίσης, προέκυψε ότι θα πρέπει ίσως να αλλάξει η χρήση των κονδυλίων και να ε, διοχετεύονται τα κονδύλια σε αυτούς που επλήγησαν σε μεγαλύτερο βαθμό από την κρίση. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόσκα. Τελευταία ομιλήτρια η κυρία Μωρίν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα συμφωνήσω απολύτως ε, με την Edith Bauer για το θέμα της επιθετικότητας και της αύξησης της βίας λόγω της κρίσης. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και θα θέλαμε και εμείς να ακούσουμε την απάντησή σας. Ε, σε σχέση με την ερώτηση για τις, για τις γυναίκες και για τα τεχνικά επαγγέλματα, ποιος επαγγελματικός προσανατολισμός υπάρχει στα σχολεία, δηλαδή ε, στους τομείς με υψηλή προσθεμένη αξία δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες, αλλά τι γίνεται ούτω ώστε ε, τα κορίτσια, τα νερά κορίτσια να μπορέσουν ε, ήδη από χαμηλή ηλικία να προσανατολιστούν προς αυτούς ε, τους τομείς με υψηλή προσθέμενη αξία, όπως μηχανική, παραδείγματο χάρη. Δηλαδή, γίνεται κάτι για να προσανατολιστούν οι γυναίκες προς αυτούς τους σταθερούς τομείς με υψηλή προσθέμενη αξία. Πρόεδρος, η κυρία Κώστα προσθέθηκε στον ε, κατάλογό μας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αλουμπράνη, για αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση που μας παρουσιάσετε και για το γεγονός ότι μας επιτρέψετε να ρίξουμε μια ματιά στα πιο γενικά και παγκόσμια θέματα. Συμφωνώ ότι το μεγάλο στίχημα αυτής της κρίσης είναι να βγούμε διαφορετικά από ό,τι εισήλθαμε και νομίζω ότι οι γυναίκες εδώ μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό και θεωρώ ότι έχουμε πάντα αυτή την υποχρέωση να βλέπουμε τις γυναίκες και ως τις πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο της ένδυας, της ε, πιο ευάλωτης κατάστασης και της ανεργίας, αλλά και ως και τα ισχυρά χαρτιά, τα στρατηγικά χαρτιά για να μπορέσουμε να εξέλθουμε από αυτή την κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αμφισημία στο θέμα των γυναικών και ίσως θα ήταν σφάλμα αν μιλούσαμε μόνο για τις γυναίκες ως θύματα και δεν ε, παίζαμε το χαρτί της επένδυσης ε, στις γυναίκες για να μπορέσουμε να εξέλθουμε με διαφορετικό τρόπο, ε, ακόμα και στο μοντέλο ανάπτυξης. Το είπατε και στο συμπέρασμά σας και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο δυσδυτικά. διότι αλλιώς η Ευρώπη και οι χώρες ε, οι αναπτυσσόμενες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ε, πρόσφατα έκανε μία έκθεση η οποία δείχνει ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή το 47% του πληθυσμού κινδυνεύει από τη φτώχεια και ξέρουμε ότι ο κίνδυνος είναι περισσότερο για τις γυναίκες για τους λόγους που μας εκθέσετε κι εσείς. Αν δούμε τα πράγματα εκτός Ευρώπης, στις αναπτυσσόμενες χώρες, ξέρουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις Υπάρχει ύφεση ε, των ανισοτήτων, υπάρχει μια αύξηση της βίας, ε, είναι πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο που μας δώσετε κι εσείς ε, σε σχέση με την οικονομική κρίση και επιπλέον υπάρχει και το θέμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ούτω καθεξής. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Εμείς θα πρέπει να δούμε και τι ακριβώς ε, μπορούμε να κάνουμε και εδώ θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και τις πιο αποτελεσματικές ε, στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας και της ανεργίας των γυναικών αλλά να κατανοήσουμε ταυτοχρόνως πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα μέτρα, τις μικροπιστώσεις και όλα αυτά τα οποία υλοποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό που άλλαξαν και τον τρόπο ε, ανάλυσης των όρων της κρίσης από πλευράς Παγκόσμιας Τράπεζας για να έχουμε ακριβώς αυτό που σας είπα, να γίνει η γυναίκα το στοιχείο δύναμης και οικονομίας. Πολλέ φορές ε, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι αν έχουμε μια μορφωμένη γυναίκα, έχουμε και παιδιά πιο μορφωμένα, γυναίκες οι οποίες δίνονται μικροπιστώσει, υπάρχουν μεγαλύτερη κύκλοι εργασία στην τοπική οικονομία και αυτό μπορούμε να κάνουμε και εμείς ως γυναίκες του δυτικού κόσμου, να παίξουμε αυτό το χαρτί. Ευχαριστώ θερμά όλους ε, τις συναδέλφους. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Λυπάμαι αλλά θα πρέπει να διακόψουμε τώρα ε, και παροτρύνοντας την κυρία Λουμπράνη όσο το δυνατόν συνταμότερα γίνεται να μας απαντήσει σε όλες αυτές ε, τις ερωτήσεις. Θα έχουμε και μελλοντικά την ευκαιρία να συζητήσουμε. Παρακαλώ κυρία Λουμπράνη. So much. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τόσο ενδιαφέρουσε αυτέ οι ερωτήσει που πραγματικά θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο να προσπαθήσω να τι απαντήσω όλε. επομένως δεν θα κάνω καμία τέτοια απόπειρα. Αυτό που θα κάνω ε, είναι το εξή. Τι έχω γράψει όλε και θα μπορούσα ίσω να σα απαντήσω γραπτό σε κάποιε από αυτέ τι ερωτήσει. Να επισημαίνω κάποια πράγματα. Σε κάποιε από τι ερωτήσει, όπω για παράδειγμα το θέμα τη βία κατά των γυναικών, ε, κατά πόσον υπάρχουν επιπτώσει ε, σε γυναίκε που ανήκουν σε μειονοτικέ ομάδε. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι όντω υπάρχει έλλειψη δεδομένων. Υπάρχει έλλειψη στοιχείων και αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερο τι ακριβώ συμβαίνει, είναι να αυξήσουμε τι επενδύσει σε αυτό και να έχουμε περισσότερα δεδομένα. Ένα από τα θέματα τα οποία θέσατε σχετίζονται περισσότερο από πλευρά λύσεων ε, στην Ευρώπη. Αυτά που κάνει η UNIFEM εστιάζει περισσότερο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το τι λοιπόν ε, αποφέρει καρπούς για να μπορέσουμε να έχουμε γυναίκες σε θέσεις εργασίας για παράδειγμα είναι αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, πρέπει όμως να συλλέξουμε και τα στοιχεία. Υπήρξαν και πολλές ερωτήσεις οι οποίες απευθύνθηκαν σε μένα. Είναι προφανώς ότι υπάρχει και μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη εδώ στην αίθουσα και εδώ πρέπει να σας πω ότι είμαστε μεν στην Επιτροπή Γυναικών αλλά υπάρχουν και άλλες επιτροπές στις οποίες οι... Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει να μαθαίνει τι συμβαίνει. Η Επιτροπή Ανάπτυξη, η Επιτροπή Περιβάλλοντο, τι συζητούν και πώ μπορείτε εσεί να συνεισφέρετε και να επηρεάσετε και τι ε, συζητήσει που γίνονται εκεί. Όχι μόνο να συζητάμε μεταξύ μα. Τώρα, σε σχέση με την ερώτηση της κυρία Ζαμπόρσκα, να πω ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν πολύ καλή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η εταιρική σχέση μπορεί να ενισχυθεί και για την ε, ατζέντα για τα θέματα ισότητας του φύλου και φυσικά το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης η οποία έγινε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο από κοινού και όχι να συνεργαζόμαστε ε, ο καθένας ξεχωριστά για κάθε θέμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια τα οποία διοχετεύονται σε μια πάρα πολύ σημαντική ε, κρίση, την ε, διατροφική κρίση. Πολλά από αυτά τα κονδύλια διοχετεύονται μέσω των Ηνωμένων Εθνών και το θέμα είναι πόσα θέματα ισότητας φύλων λήφθηκαν υπόψη εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού υπάρχουν ευκαιρίες για μας να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε. Πολλά έχουν να κάνουν με την πρόσπιση των συμφορώντων μας, κάποια είναι αλλαγές πολιτικές, πρέπει να σκεφτούμε τι στρατηγικές, πιο ακριβείς μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Όπως είπα δεν θα σας καθυστερήσω όλο, αλλά θα ρίξω μια πιο στενή ματιά για να δω αν μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένες πλήρες πληροφορίες και να δω κατά πόσο μπορεί να σας τις δώσει η Πρόεδρος από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ η κυρία Γκεμάη πολύ γρήγορα. Να κάνω μια πρόταση. Πιστεύω ότι η συζήτηση ήταν πολύ σημαντική, πολύ αποδοτική, διότι μας έδωσε το έναυσμα για να θέσουμε περισσότερο ερωτήσεις. Μήπως θα μπορούσαμε να σας καλούμε μία φορά ή δύο φορές το χρόνο, γιατί ε, έτσι θα μπορέσετε να ε, δείτε κι εσείς ότι η Επιτροπή Γυναικών θέλει να έχει μια στενότερη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κιμάη. Για άλλη μια φορά. Σα ευχαριστώ κυρία Λουμπράνη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Υπήρξαν πάρα πολλέ ερωτήσει, μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, σα ευχαριστώ πολύ και σα περιμένουμε και πάλι στην Επιτροπή. punkt på dagordningen handlar το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι προφορικές ερωτήσεις. Η ισότητα των φίλων στην εξισορρόπηση εργασίας και οικογενειακών ευθυνών. Υπάρχει μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και επιπλέον και μια πρόταση ψηφίσματος. Ο χρόνος ε, μας πιέζει σήμερα το πρωί. Ελπίζω να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τις δύο προφορικές ερωτήσεις. Αλλά ως προς το ψήφισμα και τη συζήτηση για το ψήφισμα θα επανέλθουμε στις 5 Οκτωβρίου. Θα έχουμε και το ψήφισμα στις 5 Οκτωβρίου λοιπόν και μετά θα μπορέσουμε να έχουμε και προτάσεις τροπολογίας μέχρι τις 8 Οκτωβρίου. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα μόνο τις δύο προτάσεις για προφορικές ερωτήσεις. οι διάφορες πολιτικές ομάδες ε, συμμετέχουν ε, στην εκπόνηση, στη σύνταξη αυτών των προφορικών ερωτήσεων. Νομίζω ότι ήταν πολύ υποδομητική η δουλειά μας. Να δώσω το λόγο λοιπόν για ε, τη συζήτηση. Νομίζω η κυρία Μωρίν έχει κάποια πράγματα να μας πει, διότι αυτή ασχολήθηκε με τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι για να κερδίσουμε λίγο χρόνο η προφορική ερώτηση και προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή είναι ε, αυταπόδεικτη διότι είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής ζωής και οικογενειακής ζωής ιδίως σε περίοδους κρίσεως όπως τώρα και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι θέμα θέματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί εδώ κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συγκεντρώσουν όλες τις ε, πολιτικές ομάδες ε, γύρω από αυτά τα θέματα εάν εσείς δεν έχετε αντίρρηση. Ευχαριστώ κυρία Μωρίν. Συμφωνώ με την άποψή σας ότι είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στα θέματα αυτά. και να συνδυάσουμε την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή αλλά οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να συνδυάσουν την εργασία τους με την με την οικογενειακή του ζωή και έτσι ε, ακόμη είναι το θέμα προσυζήτηση αλλά εάν κανείς άλλος δεν θέλει να λάβει το λόγο τότε θα ήθελα να παρουσιάσω να ρωτήσω συνάδελφοι εάν μπορούμε να υιοθετήσουμε τις ε, δύο προφορικές ερωτήσεις αντιλαμβάνομαι ότι μπορείτε και θέλω να ευχαριστήσω τους πάντους για την καλή αυτή δουλειά που έχουν κάνει. Τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο και πάλι είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον για την Επιτροπή μας. Πρόκειται για το πρόγραμμα της Στοκόλμης. ένα χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας. Οπότε θα έχουμε δύο αρχικές παρουσιάσεις. Καταρχήν επί των νομικών θεμάτων ε, μέσω της ε, Σουηδικής Προεδρίας, δηλαδή ο κύριος Μάγνους Γκράνερ και σε θέματα μετανάστευσης και πολιτικής ασύλου έχουμε ε, την υφυπουργό Μίντα Λιούγκρεν από την Σουηδία η οποία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Στοκόλμης. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης έχει στενή σχέση με την εργασία αυτής της Επιτροπής, ιδίω σε θέματα που έχουν ε, σχέση με τις διακρίσεις, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω τους υπουργού από την Σουηδία Λοιπόν, θα ήθελα να χαιρετήσω την κυρία Μίρνα Λιούγκρεν που είναι η πρώτη ομιλήτρια και θα εξετάσουμε την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Ε, ε, σας ε, Καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση. Είναι πολύ βασική η παρουσία σας εδώ και σας δίνω το λόγο κατευθείαν. Ε. Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε για να μιλήσουμε για το πρόγραμμα της Σουηδικής Προεδρίας, κυρίως ως προς το πρόγραμμα της Στοκχόλμης το νέο πενταετές πρόγραμμα θα αντικατεστήσει το υφιστάμενο. Είναι ένα από τα βασικότερα καθήκοντα της Σουηδικής Προεδρίας. Θα σας μιλήσω για τους γενικότερους πολιτικούς προσανατολισμούς και ο συνάδελφος μου, ο Μάγνους Γκράνερ, θα σχολιάσει τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερως την Επιτροπή σας γιατί είναι θέματα αρμοδιότητάς σας. Το νέο πρόγραμμά μας ε, για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις ε, θα είναι ένα από τα βασικότερα στρατηγικά έγγραφα ε, για τα ερχόμενα χρόνια. Η φιλοδοξία μας είναι να καταλήξουμε σε προγράμματα ώστε να έχουμε μια ασφαλέστερη, μια πιο ανοιχτή Ευρώπη όπου θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Ο βασικός στόχος είναι να είμαστε φιλόδοξοι, να έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια και να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Ισορροπημένη διότι η κοινοτική συνεργασία στον τομέα αυτό έχει αυξανόμενη σημασία τα τελευταία χρόνια. Χρειαζόμαστε ένα σαφέστερο πολιτικό πλαίσιο για να ε, υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Μακροπρόθεσμο πρέπει να είναι το πρόγραμμα, διότι θα αποτελέσει τη βάση για μια ενισχυμένη και αποτελεσματικότερη συνεργασία πέρα από τα πέντε χρόνια που θα καλύπτει αρχικά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Επίσης χρειάζεται ισορροπημένη προσέγγιση διότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα κατασταλτικά μέτρα και τα μέτρα ε, προστασίας ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα από τη σκοπιά των πολιτών. Αυτό είναι βασικός μας στόχος, ε, και θα πρέπει να καταλάβουν τη σημασία του προγράμματος οι πολίτες, ε, διότι θα προκύψουν απτά μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν και προσθέμενη αξία στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έχουν τονίσει όλα τα κράτη-μέλη σε προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε μαζί τους. Ε, οι πολίτες λοιπόν ε, θα πρέπει να ενδιαφερθούν για το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Γίνεται και στην Σουηδία μια σχετική συζήτηση και υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, υπάρχουν θελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, blog στο διαδίκτυο για αυτό το ζήτημα. Ε, και η διαδικασία μας θέλουμε να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ώστε να γνωρίζουν τι συμβαίνει οι πολίτες και να είναι πεπισμένοι ότι λαμβάνεται υπόψη η δική τους οπτική γωνία στη στοχοθέτηση του προγράμματός μας ε, αξιότιμοι βουλευτές. Ε, το φθινόπωρο θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσε συζήτησεις. Θα ακούσετε και τον συνάδελφό μου τον κύριο Γκράνερ να σε εξηγεί το πρόγραμμα μας ε, θα ήθελα απλά να αναφερθώ στις επισκέψεις που έχουν γίνει από βουλευτές του Κοινοβουλίου στην Σουηδία για τη συζήτηση αυτού του προγράμματος της Στοκχόλμης. Ε, χάρη σε όλες αυτές τις συζητήσεις μπορούμε να λάβουμε δεόντως υπόψη τις απόψεις ε, των πολιτών της Ενώσης. Από τις διμερείς επαφές που είχαμε έχω αποκομίσει την εντύπωση ότι υπάρχει μεγάλη ευρία συνένεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης. Ε, δουλειά της Προεδρίας είναι να λάβει υπόψη τις ε, απόψεις αυτές ε, κατά την εκπόνηση του προγράμματος που θα παρουσιάσουμε και θα επεξεργαστούμε κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Τέλη Οκτωβρίου η Σουηδική Προεδρία προτίθεται να παρουσιάσει το πρώτο σχέδιο του κειμένου και μετά αναμένονται εντατικέ διαπραγματεύσεις μέχρι την έγκριση του προγράμματος στη τη κορυφής το Δεκέμβριο. Ε, και για το μέλλον της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό φυσικά να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι βασικός εταίρος μας. Η Σουηδική Προεδρία επανειλημμένα έχει συναντηθεί ε, με διάφορους βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την αγαστή συνεργασία στις διάφορες συνεδριάσεις που ήδη έχουμε προγραμματίσει για το φθινόπωρο. Ε, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις δικές σας προτεραιότητες ε, για αυτό το πρόγραμμα ε, και προσβλέπουμε με ανυπομονησία στο ψήφισμα που θα εκδώσετε τον Νοέμβριο για το θέμα αυτό. Βάσει των πορισμάτων της σημερινής μας συζήτησης εδώ στο Κοινοβούλιο και βάσει της άτυπης συνεδρίας των Υπουργών στη Στοκχόλμη και βάσει των διμερών επαφών που είχαμε με τα επιμέρους μελη Η Σουηδική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το μελλοντικό πρόγραμμα της Στοκχόλμης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών. Έχουμε ένα φιλόδοξο συγκεκριμένο πρόγραμμα όπου θα ιεραρχηθούν σαφώς οι προτεραιότητες. Θεωρούμε ότι και στη συνέχεια πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή, μια διαφανή διαδικασία όπου όλα τα κράτη-μέλη, όλα τα θεσμικά όργανα, όλοι οι εταίροι κλειδιά θα συμμετάσχουν ενεργά. Ε, και ε, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα αποτελέσει βάση και για μελλοντικές εργασίες ε, και το φθινόπωρο θα γίνουν πάρα πολλές επικοδομητικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δική σας δράση θα έχει καταλητικό χαρακτήρα για το τελικό αποτέλεσμα. Ε, πρέπει να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα ε, για το οποίο θα υπάρχει ευρεία υποστήριξη από πλευράς κρατών μελών και από πλευράς ε, θεσμικών οργάνων της Ένωσης, μεταξύ των οποίων και το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τώρα θα δώσω το λόγο στον Μάγνους Γκράνερ. Υφυπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προεδρέ αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Γυναικών. Έχουμε γενικούς στόχους ε, στη Σουηδική Προεδρία. Ένας από αυτού είναι να αυξήσουμε την ασφάλεια ε, και την προστασία των πολιτών της ευρωπαϊκή Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος της Στοκχόλμης. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδώσει μία ανακοίνωση που κατά τη γνώμη μας έχει κεντρικό ρόλο για να ληφθούν υπόψη τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σεβασμός, παραδείγματος χάρη της νομοθεσίας για την κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης. Αυτό καλύπτει όλες τις μορφές διακριτικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας, λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ε, πεπιθήσεων, ε, θρησκείας, ε, αναπηριών. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να ρίξουμε βάρος είναι τα μέτρα που χρειάζονται ούτω ώστε να έχουμε αυξημένη ε, προστασία για τα ε, άτομα που ε, όπως οι γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία που υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Η προστασία των θυμάτων είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες στο μελλοντικό πρόγραμμα. Το να είναι κανείς θύμα προκαλεί συχνά τραύματα στη ζωή του ανθρώπου και, ε, όταν, και κυρίως όταν ε, υφίσταται κάποιος ένα, ε, μια αξιόπινη πράξη, ένα έγκλημα σε μια άλλη χώρα. και ε, αυξάνεται ορισμένες φορές ο κίνδυνος του να υποστεί κάποιος σε μια εγκληματική πράξη όταν ταξιδεύει σε άλλες χώρες και γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρει ο κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενημερώνεται και θα προστατεύεται δεόντως ε, ε, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό το θέμα έχει τονιστεί ως προτεραιότητα στο παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα θέλαμε να υπολογίζουμε στη δική σας υποστήριξη και στην επικοδομητική συνεργασία για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων ε, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πολέμηση τώρα της εμπορίας ανθρώπων. Άλλη μια προτεραιότητα της Σουηδικής Προεδρίας. Ε, τα ευπαθή ε, άτομα, οι γυναίκες, ε, τα παιδιά, η προστασία τους κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και άλλων αξιόπινων πράξεων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί σε σαφή προτεραιότητα. Υπάρχει και διεθνή συνεργασία που αποτελεί εκ των όνου για να επιτύχουν οι κοινοτικέ μας προσπάθειες. Φυσικά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο Συμβούλιο η οδηγία για την εμπορία ε, ανθρώπων και ελπίζουμε να εγκριθεί μέχρι το τέλος ε, του τρέχοντος. Η απόφαση η πλαίσιο αυτή ε, θα είναι ένα βασικό εργαλείο για την κοινοτική συνεργασία στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. Αλλά δεν παρκεί η κοινή δράση, η κοινοτική πρωτοβουλία στον τομέα αυτό γιατί υπάρχουν και οι τρίτες χώρες, οι χώρες προέλευσης, οι χώρες διαμετακόμισης, ε, συγγνώμη, διέλευσης που πρέπει να συνεργαστούν συνεργαστούν μαζί μας ε, για να επιτύχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η Σουηδική Προεδρία αποφάσισε να αναδείξει ύψιστη προτεραιότητα αυτό το θέμα στις διμερείς επαφές που έχει με τρίτες χώρες και επίση ε, θα διοργανώσουμε ε, μία διυπουργική διεθνή διάσκεψη για το θέμα αυτό στις 19 και 20 Οκτωβρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά θα προσκληθεί στην διάσκεψη που θα γίνει τον Οκτώβρη ε, και ε, αναμένουμε αθρώα προσέλευση από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Ε, ευελπιστούμε ότι η διάσκεψη θα οδηγήσει σε ανταλλαγή απόψεων και των πρακτικών στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να εγκριθεί ένα action-oriented paper, ένα έγγραφο δηλαδή πολιτικής που θα λειτουργήσει ως κατευθυντήρια γραμμή για τη μελλοντική μας δράση στον τομέα αυτό. Οφείλουμε επίσης να ενισχύσουμε την διασυνοριακή ευρωπαϊκή συνεργασία για την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας των ανθρώπων. Το θέμα της εμπορίας ε, των ανθρώπων ε, είναι πάρα πολύ επίκαιρο, πολύ πιο επίκαιρο το 2009 σε σχέση με ε, προηγούμενα χρόνια. Το Σεπτέμβριο έγινε ένας πρώτος γύρος συζητήσεων και τονίστηκε η σημασία του ζητήματος και τονίστηκε η ανάγκη ανάληψης ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση του φαινομένου. Φυσικά θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το ζήτημα από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Από πλευρά ειδικής Προεδρίας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε το πρόγραμμα της Στοκχόλης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στι επιθυμίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε φυσικά να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και ήδη είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις για την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και είμαι πλήρως πεπισμένη ότι οι συνάδελφοι έχουν ερωτήσεις ε, και επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ε, δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Χιμένης Βεζερίλ. Και σας ενημερώνω ότι πρόκειται για θέμα που είναι αντικείμενο συνεργασίας διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου. Έχουμε την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών που συνεργάζεται μαζί μας, την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Άσκο όπως ονομάζεται. Υπάρχει λοιπόν ε, συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες συναρμόδιες επιτροπές. Θα δώσω το λόγο τώρα στην εισηγήτριά μας, ε, η κυρία Χιμένες. Έχει το λόγο, παρακαλώ. Sí, <clears throat> eh, Καλημέρα, κυρία Γκρένερ, κύριε, Γκρένερ, κυρία Λούγκρεν. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω κυρίως τον ε, κύριο Γκράνερ, όταν μιλάτε για ευρωπαϊκή συνεργασία για την προστασία των θυμάτων βίας, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον ε, Έχετε κάποια ιδέα για το κατά πόσον μπορεί να προχωρήσει αυτό επί Σουηδικής Προεδρίας ή μπορεί να το προχωρήσει ιδιαίτερα η Ισπανία, αν μπορείτε να το ξεκινήσετε εσείς, να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προστασίας των Θυμάτων. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύεται μια γυναίκα στην Ισπανία όταν θα πάει και όταν φύγει να πάει στην Αγγλία ή στην Γαλλία να συνεχίσει να προστατεύεται. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να απαντάτε σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά για να είναι σαφής και συγκεκριμένη η απάντηση που δίνετε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο ο κύριος Γκράνερ. Αρχικά θα έλεγα ότι ε, δυστυχώς το ζήτημα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων ε, δεν πρόκειται να βρει την οριστική λύση του μέσα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Δυστυχώς είμαι επιπισμένος ότι το ζήτημα αυτό απασχολεί ε, όλους τους πολιτικούς της Ευρώπης και θα μας απασχολεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς θα επομιστούμε το δικό μας, τη δική μας ευθύνη στα πλαίσια του προγράμματος Στοκχόλμης, αλλά δείτε και τη θετική πλευρά, δηλαδή υπάρχει ε, ε, μια ευρεία συσπήρωση, αν θέλετε, συνένεση σχετικά με την σημασία που έχει το ζήτημα της προστασίας των θυμάτων. Ε, δείτε, πέρα από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, αναμένουμε και μία πρόταση αναθεώρησης υφιστάμενων νομικών εργαλείων δεν ξέρουμε ακριβώς ε, ποια θα είναι η σχέση ανάμεσα στην αναθεώρηση αυτών των νομοθετημάτων ε, και το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Δεν μπορώ να επισέλθω προς το παρόν σε λεπτομέρειες, ε, αλλά θα πρέπει να γίνουν και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πράγματα για την καταπολέμηση του φαινομένου. Ε, πρόεδρος, έχω δει πολλά μέλη στον κατάλογο των ομιλητών. Βλέπουμε ω εκ τούτου πόση μεγάλη σημασία έχει το ζήτημα για τα μέλη τη επιτροπή μας. Ε, ε, ε, κυρία Παπαδοπούλου. Thank you very much, Mrs. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε και η ερώτησή μου είναι για τον κύριο Γκρούνερ. Διάβασα το πρόγραμμα και όντως είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Υπάρχουν ε, κάποιες αναφοράς ε, στην ε, ποιότητα των φύλων και κατά την άποψή μου υπάρχει μία νοοτροπία ότι τα... οι γυναίκες είναι θύματα διότι μιλάμε για την ανάγκη να προστατεύσουμε τις γυναίκες από τη βία, από το δουλεμπόριο, από τις τρομοκρατικές πράξεις, από τη βία στο σπίτι και όλα ε, αυτά είναι μορφές βίας κατά των γυναικών. Η ερώτησή μου είναι γιατί δεν ε, συμπεριλαμβάνεται και κάποια μέτρα ενδυνάμωσης για τις γυναίκες στο πρόγραμμα. Διότι οι γυναίκες ε, σήμερα διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή, στον πολιτιστικό τομέα, σε όλους τους τομείς της ζωής και εμένα θα με βοηθούσε να δω ότι στο επόμενο, στα επόμενα πέντε χρόνια το πρόγραμμα αυτό θα δώσει τα μέσα στις γυναίκες να είναι πιο δραστήριες στην πολιτικό βίο, διότι ξέρουμε ότι η εκπροσώπηση σε διάφορες θέσεις ε, λήψης πολιτικών αποφάσεων είναι ε, χαμηλή και υπάρχει έλλειμμα γυναικών. Αντί λοιπόν να παρουσιάζουμε τις γυναίκες μόνο ως θύματα, θα ήθελα να σας ζητήσω και για περισσότερα μέτρα να ενθαρρύνετε τις γυναίκες να αποδείξουν την αξία τους, ώστε να μπορέσει να επιφαληθεί και η κοινωνία από τον ενεργό τους ρόλο ε, για να οικοδομηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τους ε, ανθρώπους. Τι έχετε να πείτε από αυτό. Σας ευχαριστώ. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Γκράνερ που θέλει να απαντήσει. Συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Γενικότερα οι γυναίκες δεν είναι θύματα. Ο στόχος εδώ είναι να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες, ε, να τονίσουμε τη σημασία του empowerment ε, στο οποίο αναφερθήκατε. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι συνίσταται το πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα αυτό ε, καλύπτει τα ζητήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Δεν φέρει γενικώ επί της κοινωνίας. Ε, μιλάμε για τις αρχές επιβολής ε, νόμου και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν. Μιλάμε για το νομικό πλαίσιο της δράσης τους. Δυστυχώς, η... στο στην ομάδα των θυμάτων υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες, ας το πούμε έτσι, για διάφορα, ε, για διάφορα είδη βία, στα εγκλήματα τιμής παραδείγματος χάρη. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να χειριστούμε το θέμα από πλευρά ε, των αστυνομικών αρχών μεταξύ άλλων. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι πιστεύουμε ότι γενικότερα είναι θύματα οι γυναίκε μέσα στην κοινωνία. Ε, καμία Σουηδέζα θα, δεν θα πίστευε ότι αυτό μπορεί να είναι η βάση του προγραμματός μας, αυτή η αντίληψη.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 Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Είναι πολύ ε, χρήσιμο και όντως ε, είναι βασικό να μπορούμε να προωθήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και να αποφεύγουμε την σωματεμπορία. Ξέρουμε όμως ότι η Δανία έχει εδώ μία επιφύλαξη στον τομέα αυτό. Οπότε θα θέλαμε να ξέρουμε ε, τι γίνεται. Ε, ε, στο, θέμα ασύλου και μετανάστευσης ε, η, η μετανάστευση η οποία είναι πολύ περιορισμένη αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να αναπτυχθεί και εδώ σκέφτομαι τις συζητήσεις τις οποίες έχετε οργανώσει με τα κράτη-μέλη και όπου είπατε ότι υπάρχουν ε, διμερείς ε, διαπραγματεύσεις μήνα οπότε τι γίνεται σχετικά με την πολιτική μετανάστευση τι θα πρέπει να αναμένουμε κατόπιν αυτών των συζητήσεων. Ευχαριστούμε κυρία Τόμσεν. Ε, στρέφομαι προς την Μίνα Γιούγκριεν ε, για να απαντήσει στο ερώτημα για το θέμα της ε, πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Για το κοινό σύστημα ασύλου ήδη τρέχουν διάφορα προγράμματα, έχει χαραχθεί μία γραμμή μέχρι το 2010 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προσπάθειές μας ε, για την κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Υπάρχουν επίσης ε, διάφορα ε, νομοθετήματα που εξετάζονται αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε ότι θα εγκριθούν σύντομα, κυρίως ε, αυτό που αφορά το, την ε, κοινή υπηρεσία στήριξης. Ε, ελπίζουμε να εγκριθούν υπό Σουηδικής Προεδρίας. Συνεχίζουμε λοιπόν να ακολουθούμε την πολιτική που έχουμε προσδιορίσει στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης και συνδυασμό με αυτό ελπιστούμε να εγκριθεί και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Στις διμερείς επαφές που κάναμε τα κράτη-μέλη το Σεπτέμβριο δεν μπορέσαμε ακόμη να δώσουμε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του προγράμματος Στοκχόλμης, αλλά η γενικότερη εντύπωση, όπως είπε και ο συνάδελφος μου, ο κύριος Μάγνους Γκράνερε, ε, η γενικότερη εντύπωσή μα είναι ότι υπάρχει μια συσπήρωση, μια συνένεση για τις βασικές γραμμέ του προγράμματος και μία από τις κοινέ γραμμέ είναι η πολιτική της, ε, του ασύλου και της μετανάστευσης. Τα κοινά εξωτερικά σύνορα ε, καθιστούν αναγκαίους του κοινού κανόνες για τα θέματα αυτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τόμσον. Δεν αναφέρθηκα στην πολιτική ασύλου, αλλά αναφέρθηκα στην ε, πολιτική μετανάστευσης. Για την παράνομη μετανάστευση φαντάζομαι μιλάτε. Ε, στο τομέα αυτό Οι σχετικές οδηγίες, η τροποποίηση προηγούμενων οδηγιών μας ε, δείχνουν ότι στα κράτη-μέλη, σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει φιλοδοξία να σημειωθεί πρόοδος, περαιτέρω πρόοδος σε αυτό το τομέα. Βέβαια, ε, λόγω της οικονομικής κατάστασης επιβραδύνεται η διαδικασία. Πάντως, Ε, το Δεκέμβριο άρχισε να ισχύει μια νέα νομοθεσία στο, στην αγορά εργασίας ε, για τους μετανάστες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ω βάση για τις μελλοντικέ εργασίες αλλά σε κοινοτικό επίπεδο. θα πρέπει να δούμε ε, για ποια πράγματα μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Πάντως συνεχίζονται οι εργασίες μας και οι οδηγίες ε, που ε, συζητιόντουσαν ε, έχουν παγώσει κάπως και περιμένουμε περαιτέρω πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να κάνω εγώ μία ερώτηση για την μετανάστευση για λόγους εργασίας ε, και τη μετανάστευση γενικότερα. Υπάρχουν διατάξεις για την μπλε κάρτα που μπορείτε να σχολιάσετε. Γενικότερα για την μετανάστευση είπατε ότι έχουν παγώσει λίγο οι οδηγίες ε, γιατί δεν υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον και αναρωτιέμαι, είναι λόγω της κρίσης, τι ακριβώς ε, συνέβη ε, και έχει σε τέλμα η κατάσταση, γιατί δεν σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση. Εγώ θα ήθελα να μάθω σε τι οφείλεται αυτό. Επίσης, και ο κύριος Γκράνερ και εσείς ε, είπατε ότι ε, το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμη συμπεριλαμβάνει και την συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Για την μεταναστευτική πολιτική λοιπόν, Ποια συνεργασία υπάρχει με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με διεθνεί οργανισμού κτλ. Κάτι άλλο τώρα. Το πρόγραμμα τη Στοχόλμη θα έχει σοβαρό αντίκτυπο, παραδείγματο χάρη για τι ελευθερίε των πολιτών, την ε, ε, ε, κυριότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι ζητήματα που μας καίνε εδώ στην Επιτροπή. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τη συνεργασία που ήδη υπάρχει με άλλους οργανισμούς ώστε να κατοχυρώσουμε, να διαφυλάξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ακαιρεότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια χάρη σε αυτό το πρόγραμμα. Παρακαλώ. Θα αρχίσω με τις ερωτήσεις ε, που μου απευθύνατε σε μένα και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκράνερ. Ε, με ρωτήσατε ποιος είναι ο λόγος καθυστέρησης ε, των εργασιών για την μετανάστευση, για εργασιακούς λόγους ή γενικότερα για την μετανάστευση. Καλύτερα να απευθύνετε αυτά τα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εγώ μόνο να υποθέσω μπορώ το λόγο. Και τεκμέρο ότι οφείλεται στην οικονομική δυσπραγία ε, η καθυστέρηση που δεν αφορά μόνο την Ευρώπη αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω αυτό είναι ένας λόγος που καθυστερεί τις εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευση για λόγους εργασίας. Ε, σχετικά τώρα με τους οργανισμούς με τους οποίους ε, συνεργαζόμαστε, ε, UNHCR παραδείγματος χάρη από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι ένας επιθανός εταίρος. Μπορούν ε, στον οργανισμό αυτό του ΟΗΕ να ε, συνεργαστούν με το νέο υποσύσταση γραφείο στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που τώρα μου διαφεύγουν, ε, δεν μπορώ να τους κατονομάσω, αλλά θα υπάρξει ευρεία διεθνή συνεργασία. Μάγνους, ναι, να προσθέσω και εγώ κάτι για να είναι πλήρης η απάντηση. Μπορούμε να πούμε ότι για το μέλλον Έχουμε το σχέδιο ε, τη τη στο Στοχόλμης που συζητείται εδώ και δύο χρόνια. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, περνάει από την διαδικασία εξέβρεσης συνένεσης. Ε, δεν θυμάμαι ε, αν 700 900 απαντήσεις από τη ε, διαβούλευση ε, που οργανώσαμε από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από διάφορους οργανισμούς, agencies στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από κρατικές αρχές, Έγινε πάρα πολύ, με σουηδικό τρόπο η διαβούλευση, πολύ ανοιχτή, πολύ διαφανής και ο Γενικός Διευθυντής ε, του Οργανισμού ε, Προστασίας ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι βασικός εταίρος στη διαδικασία συναντήθηκε μαζί μου σήμερα τον πρωί όταν ερχόμουν στο Κοινοβούλιο και μου είπε ότι θα τοποθετηθεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις απόψεις του. Σε αυτή τη διαδικασία είναι σαφές ε, ότι ό, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη το Σεπτέμβριο σε επαφές που είχαμε μαζί τους ε, ρίχνουν το βάρος στις ανάγκες ε, των ανθρώπων, στα δικαιώματα των πολιτών, ε, στην προστασία που χρειάζεται. Αυτό είναι πυρήνα των συζητήσεων που γίνονται με τα κράτη-μέλη. Οπωσδήποτε πρέπει να αποτελέσει αυτό το σημείο κλειδί του προγράμματος Στοκχόλμης και η προστασία των πολιτών. Ένα θέμα πολυδιάστατο, μία από τις τονίστηκε στο πρόγραμμα της σε προστασία ε, κατά των επιθέσεων, τρομοκρατικών επιθέσεων, ε, οργανωμένου εγκλήματος. Ε, κάτι άλλο που θα τονιστεί στο πρόγραμμα τη Στοχόλμη είναι η προστασία τη ανθρώπινη ακαιρεότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που θέτουν. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Γκράν και την κυρία Γιόγκριν για τις παρουσιάσεις τους. Δώσατε σαφέστα τις απαντήσεις και... Ε, ξέρω ότι είσαστε πάρα πολύ αποσχολημένοι και πρέπει να αποχωρήσετε τώρα γιατί πήγε ώρα 11.30. Πάντως σας ευχαριστούμε που ήρθατε και προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ε, Προτείνω να συνεχίσουμε με την ημερήσια διαταξή μας. Τώρα θα συζητήσουμε την έκθεση της κυρίας Χιμένες, της κυρίας Χιμένες Μπεσερίλ, που είναι η συγγήτριά μας. Σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ναι, καλημέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να σας παρουσιαστώ για όσους δεν με γνωρίζουν. Λέγομαι Τερέσα Χιμένεθ Μπεθερίλ και όποιος ρωτήσει στη χώρα μου για μένα ή ψάξει να με βρει, το όνομά μου σχετίζεται πάντα με την προάσπιση της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης. Αυτό που έκανα δηλαδή τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ήταν η προάσπιση των θυμάτων, πιο συγκεκριμένα των θυμάτων ε, τρομοκρατίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έκανα μόνο αυτό. Προάσπισα πάντα ε, θύματα τα οποία ε, όπως ανακάλυψα εγώ ε, ασχολούμενοι πάντα με τα θύματα και εργαζόμενοι πάντα μαζί τους από όπου και να προέρχονται από ποιο λόγο και να έχει προκύψει ε, το γεγονός ότι είναι θύματα ε, αναζητούν τη δικαιοσύνη. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και λοιπόν και να ευχαριστήσω την Επιτροπή αυτή που μου επέτρεψε να εκπονήσω αυτό το ψήφισμα ε, για το πρόγραμμα της Στοχόλμης που αναφέρεται ακριβώς ε, σε αυτό το οποίο εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, η αναζήτηση της ασφάλειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να εκθέσουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση είναι μια σειρά από σημεία προκειμένου να δώσουμε μια όθηση για κάτι το οποίο θεωρώ ότι λείπει από το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τη γυναίκα, πριν έλεγε και μια συνάδελφος, ότι ούτε και σε μένα να αρέσει να είναι θύμα, σε κανέναν δεν αρέσει να είναι θύμα και οι γυναίκες δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται πάντα ω θύματα σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν μπορούμε επίσης να αρνηθούμε ότι εξακολουθεί να υφίσταται μια κατάσταση στην οποία η γυναίκα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση όταν έχουμε περιστατικά βία, ε, σωματεμπορία, τρομοκρατία, η περίπτωση, η θέση της γυναίκας είναι πολύ πιο ευάλωτη και βρίσκεται πάντα ανανεμιγμένη σε αυτές τις υποθέσεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που το αντικατοπτρίζει αυτό το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Στο πρώτο σημείο το οποίο έχετε θα δείτε ότι ε, υπάρχει μία παρακίνηση προς το Συμβούλιο για να εμείνουμε στα θύματα ε, βίας και γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τόσο η Σουηδική αλλά και η Ισπανική ε, Προεδρία να προχωρήσει αυτό το ένταλμα για τα ε, θύματα και θεωρώ ότι επιμένω τα θύματα θα πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις χώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν το επιτύχουμε αυτό, παρά το γεγονός ότι θα είναι δύσκολο, ε, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να πολεμήσουμε, θα ήταν πολύ σημαντικό. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι τα θύματα τρομοκρατίας είναι και έμεσα θύματα. Δεν υπάρχουν μόνο τα άμεσα θύματα, αλλά υπάρχουν και τα έμεσα θύματα στην πλειονότητά του μητέρε, γυναίκε, χείρε. Δεν αναφερόμαστε σε αυτέ, αλλά εγώ που κινούμαι μεταξύ των θυμάτων πρέπει να σα ε, διασφαλίσω ότι όποιο ε, θέλει να προχωρήσει, θέλει να διαφυλάξει τα παιδιά του, να διαφυλάξει την οικογένειά του και που κάθε μέρα μάχεται για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια και για όλες αυτές τις αξίες ε, που είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι οι γυναίκες. Και όταν ε, ε, μιλάμε με οργανώσεις θυμάτων τρομοκρατίας όπως αυτό στο Παρίσι για παράδειγμα είχαν κόσμο από, την, από το Ισραήλ, από την Ιρλανδία, από τη Ζιμπάμπου, από όλες τις χώρες. Το 90% είναι γυναίκες. Από την Ισπανία όλες είναι διαφορετικές. Η κάθε μία με ένα ιστορικό τελείως διαφορετικό, αλλά όλες αυτές έχουν ένα κοινό αγώνα και είναι γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει κάποια μνήα σε αυτή την αξία των γυναικών και στο πόσο ε, πάσχουν αυτές οι γυναίκες ως έμεσα θύματα της τρομοκρατίας. Στο τρίτο σημείο Επισημάνεται ο ρόλο που διαδραμάτισε το πρόγραμμα Δάμφνη στο πρόγραμμα της Στοχόλμη. Ε, θέλει να προσφέρει πάντα μεγαλύτερη προστασία στις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Και φυσικά ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προχωρήσει η Ισπανική Προεδρία. Εδώ, μιλώντα για τα θύματα, ήθελα να πω και κάτι το οποίο δεν είπα ίσω στο σημείο 1, είναι η σημασία των νέων θυμάτων. Δεν ξέρω τι γίνεται στη χώρα σα, αλλά στη χώρα μου υπάρχει μια τεράστια αύξηση δολοφονιών ε, κοριτσιών 17-16 ετών, ανήλικες, αλλά είναι γυναίκες. Πολλές φορές βιάζονται και κατόπιν δολοφολούνται και ε, συνήθως είναι άνθρωποι στον στενό τους περίγυρο. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι κοπέλες να προστατεύονται. Τώρα, μιλώντας για βία στο σπίτι, θα ήθελα να σταθώ σε μία έκθεση του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει ότι η βασική αιτία θανάτου γυναίκων, γυναικών μεταξύ 19 και 40 ετών πέραν του καρκίνου και των ε, αυτοκινητιστικών ε, ατυχημάτων είναι η βία στο σπίτι. Επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία αυτά και να πολεμήσουμε γι' αυτό. Θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε και για τις γυναίκες μετανάστριες. Εγώ που ζω μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας διαπίστωσα ότι υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις στην ε, Ιταλία. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια Ιταλίδα συνάδελφος εδώ που μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση. Υπάρχουν ε, κοπέλες μετανάστριες που είναι Ευρωπαίες, διότι ούτως ή άλλως ε, ζουν πάρα πολλά χρόνια, πηγαίνουν σχολείο στις χώρες μας, στην Γαλλία, στην Αγγλία αλλά μετά στην οικογένεια εξακολουθούν να ζουν με αυτή τη βία. Η βία μπορεί να προέρχεται από τον πατέρα τους. Σε μια περίπτωση που είχαμε στην Ιταλία είχαμε πάρα πολλούς ε, θανάτους ε, από τον πατέρα ή από το φίλο τους ή από ανθρώπους στο στενό τους ε, οικογενειακό κύκλο. Ε, από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης λοιπόν εμείς ως Επιτροπή Γυναικών θα έπρεπε να ζητήσουμε την προάσπιση αυτών των Ευρωπαίων ε, γυναικών, είτε προέρχονται από το Μαρόκο, είτε προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αυτές θεωρούν ότι είναι Ευρωπαίες και θέλουν να ζήσουν όπως εμείς. Επομένως, δεν μπορούμε να τις αφήσουμε προστάτευτες. Τέλος, ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για αυτό που είπε ο κύριος Γκράνερ, που είναι ε, το σύγχρονο δουλεμπόριο. Θεωρώ ότι είναι θεμελιώδες δεν θα αρκεί μόνο μία δικαστική απόφαση, αλλά να συνεχίσει να υπάρχει και βοήθεια ψυχολογική, μια δυνατότητα ένταξης, ώστε όλα αυτά τα άτομα που θέλουν να συνεργαστούν και συνεργάζονται να μην βρεθούν στο περιθώριο κατόπιν της δικαστικής απόφασης, να μπορέσουν να επανενταχθούν στην εργασιακή ζωή και να έχουν μια ζωή χωρίς φόβο, να μην ζουν με το φόβο, ε, διότι μπορεί να ζουν όλοι τους τη ζωή με φόβο. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν και την άποψή σας. Εγώ ήθελα να διευκρινίσω απλά λίγα πράγματα στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συγγήτριά μας έχει πάρα πολλές γνώσεις και είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη και προσιλωμένη στη δουλειά της. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Έχω διαβάσει φυσικά το ψήφισμα και άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την παρουσίαση. Βλέπω ποια είναι τα σημαντικά σημεία, όλα συμπεριλαμβάνονται μέσα στο ψήφισμα και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συσπηρωθούμε γύρω από το ψήφισμα και να υποστηρίξουμε ε, την πλειοψηφία των σημείων που καλύπτεται. Απλά για το σημείο 5 θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μιλάτε για την εμπορία των ανθρώπων. Είναι ε, ε, αυτό συνεπάγεται ένα πελώριο πρόβλημα για την κοινωνία μας και θεωρώ ότι κάτι λείπει εδώ. Δεν μιλάμε για την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικούς ε, σκοπούς, δηλαδή για το σκοπό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Υπάρχουν πάρα πολλά αριθμητικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι αυτός είναι ένας από, ο βασικότερος στόχος ε, της εμπορίας ανθρώπων, η σεξουαλική ε, εκμετάλλευση. Οπότε, μήπως θα έπρεπε να προσθέσουμε κάτι σχετικό μέσα στο ψήφισμα για να είναι πληρέστερο. Κατά τα λοιπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Κώστα μας έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της. και να τη συγχαρώ και για τις αρμοδιότητές της. Ε, κάποιες σκέψεις. Η πρώτη μου είναι η εξής. Μήπως σε σχέση όλου του με όλο το πρόγραμμα της Στοχόλμης, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά σημεία, ίσως θα μπορούσαμε, επιτρέψτε μου να σας το προτείνω, ίσως και ως προήμιο, ένα κείμενο εντός εισαγωγικών από πλευράς φύλου, το οποίο θα αξιολογεί ε, λίγο ευρύτερα το ρόλο των γυναικών σε όλη τη στρατηγική. Η στρατηγική αφορά κυρίως ε, την εμπορία ανθρώπων, τη βία κατά των γυναικών, αλλά να έχουμε μια ευρύτερη λίγο έννοια, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά που έλεγε και πριν η κυρία Παπαδοπούλου, όχι να ξεχνάμε τα θύματα, αλλά να πούμε ότι σε όλη τη στρατηγική της Στοκόλμης θα πρέπει να δοθεί ε, μια κάποια υποστήριξη και να γνωστοποιηθεί και όλο το θέμα αυτών των γυναικών που δεσμεύονται και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στη ποινική δομή και που συνήθως είναι το πρώτο ε, όριο αν θέλετε. Πάρα πολλές γυναίκες για παράδειγμα στην αστυνομία έχουν αφιερωθεί στην βοήθεια των γυναικών που είναι θύματα. Υπάρχει δηλαδή ε, και όλο αυτό το θέμα που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοχόλμης. Ε, υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία συμμερίζομαι στην ε, γνωμοδότηση της κυρίας Χιμένες και, Χιμένες και εγώ θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να μιλάμε και επίσης εμπόριο ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και εργασιακή εκμετάλλευση. Θα ήθελα επίσης στη γνωμοδότηση πέραν των νέων γυναικών να μιλάμε και για αναλύκου εν γέννη, διότι είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε ε, ιδιαίτερη προσοχή και συμφωνώ απόλυτα με το θέμα των έμεσων θυμάτων. Έχουμε μια συνάδελφο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Μπορσελίνο, η οποία είναι έμεσο θύμα, αδερφή του δικαστή που δολοφονήθηκε και αυτή από αυτή την αδυναμία, αδυναμία της ε, ε, εκμεταλλεύτηκε θετικά την κατάσταση, πηγαίνει στα σχολεία και μιλά για την κατάσταση στην Ιταλία. Τρεις πιθανές προτάσεις τώρα. Το πρώτον, όταν ε, μιλάμε για την υποστήριξη της κυβέρνησης. Λέμε γυναίκες μόνες χωρίς ε, ε, υποστήριξη της ε, κυβέρνησης. Ε, και υπάρχει όμως και μία αποζημίωση, για παράδειγμα. Υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες. Εμείς στην Ιταλία έχουμε νομοθεσία για αποζημίωση. αν έχουμε λοιπόν και αυτή τη συνδρομή πέραν φυσικά της ψυχολογικής και λοιπά υποστήριξης. Τώρα, ε, ανηλίκους να τους συμπεριλάβουμε στο σημείο για το πρόγραμμα Δάφνη, γιατί το πρόγραμμα Δάφνη αφορά και ανήλικα άτομα και όχι μόνο γυναίκες και το τρίτο σημείο, εξ όσων γνωρίζω εγώ, αλλά μπορείτε να είστε πιο ενημερωμένοι, τα περιστατικά βία στο σπίτι είναι ο η πρώτη αιτία θνησιμότητας και μέσα σε αυτό έχουμε και τη βία στο σπίτι. Δεν νομίζω ότι η βία σαν βία στο σπίτι, αλλά τα ατυχήματα εντός του σπιτιού. Αλλά φυσικά είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και είναι σε αύξηση. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να το διευκρινίσουμε, να το επαληθεύσετε κιόλα, διότι μπορεί να είναι και υπερβολή να λέμε κάτι τέτοιο και να το παρουσιάζουμε εδώ στατιστικό στοιχείο. Τώρα, το θέμα του ρόλου των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εγώ θα ήθελα να επισημάνουμε ίσως λίγο περισσότερο την υποστήριξη των κυβερνήσεων και το ρόλο που οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πολλές γυναίκες στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις κάνουν για το εμπόριο ανθρώπων. Ε, και επίσης να επισημάνουμε και τη στενή σχέση μεταξύ μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων και τοπικών αρχών, οι οποίες κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για την επανένταξη. Και επειδή εκεί η παρουσία των γυναικών είναι πολύ σημαντική και είναι οι πλέον αρμόδιες, θα πρέπει να έχουμε και μια θετική επισήμανση από αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κώστα. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. μπορείτε να σχολιάσετε ε, την συζήτηση που κάναμε ή μπορείτε να διευκρινίσετε διάφορα σημεία από, ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση από τους δύο υφυπουργούς που είχαμε νωρίτερα. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ίσως ε, μπορώ να διευκρινίσω αυτό το οποίο ελέγχθη σχετικά με την νόμιμη μετανάστευση και την ε, ε, νομοθετική διεύρυνση διότι για να τοποθετήσω τα θέματα μέσα στο πλαίσιο τους είχαμε προβλήματα νομοθετικά για δύο λόγους. Καταρχήν διότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο χώρο, ιδίω για ορισμένα κράτη-μέλη και δεύτερον διότι πρέπει να θυμίσουμε ότι ο μηχανισμός της νομικής βάσης προβλέπει την ε, ομόφωνη ε, υιοθέτηση από το Συμβούλιο. Πράγμα το οποίο καθιστά πολύ δύσκολο το θέμα, διότι το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει μία πρόταση για την ε, πρόσβαση στην αγορά εργασίας που απεσήρθη διότι μπλόκαρε. Μετά υποβάλαμε μία πράσινη βίβλο, ένα πρόγραμμα δράσης και τώρα μία πρόταση σχετικά με την μπλε κάρτα η οποία έχει υιοθετηθεί και έχει μπλοκάρει μια άλλη πρόταση στο Συμβούλιο για την ε, ενιαία άδεια και αυτό πρέπει να ε, ισχύσει τουλάχιστον για τους ε, μετανάστες οι οποίοι εργάζονται νόμιμα στην κοινότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διέξοδο λόγω των αντιδράσεων ορισμένων κρατών μελών, της δύσκολης κατάστασης της αγοράς εργασίας που δεν διευκολύνει άλλωστε τα πράγματα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει δύο ακόμη προτάσεις που αναφέρεται τους εποχικούς εργαζομένους και για τις μεγάλες επιχειρήσεις και οι προτάσεις αυτές θα παρουσιαστούν εντός των επόμενων μηνών. Σχετικά με το πρόγραμμα της Στοχόλμης για την νόμιμη μετανάστευση θέλουμε να βελτιώσουμε και να ανασκευάσουμε τα ισχύοντα κείμενα και όσον αφορά την επανένωση των οικογενειών θα πρέπει να υπάρξει μία πρόταση αλλαγής η, εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας οπότε από μηχανισμό απόφασης περνάμε σε συναπόφαση και όπου θα υπάρξει μεγαλύτερη δυναμική στις διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δεν έχω συγκεκριμένες προτάσεις Προφανώς το πρόγραμμα της Στοχόλμης που καλύπτει λίγο πολύ όλη την ε, ε, δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις ήμασταν προσεκτικοί και η Επιτροπή χαιρετίζει οποιαδήποτε πρόταση ε, μπορεί να βελτιώσει την πτυχή που αναφέρεται στις γυναίκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτές τις διευκρινήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο κύριος Μενές θέλει να προσθέσει κάτι, η κυρία Χιμένες θέλει να προσθέσει κάτι για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ναι, να ευχαριστήσω την κυρία Κώστα για όλα τα στοιχεία που μας έδωσε και εσάς κυρία Πρόεδρε. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που θα κάνω τώρα είναι να τα δω όλα αυτά, να προτείνουμε τροπολογίες και εγώ θα κάνω κάποιες αλλαγές. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους ε, να έχουμε τροπολογίες προκειμένου να βελτιώσουμε το κείμενο αυτό και ελπίζω από το κείμενο αυτό να προκύψει κάτι το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει στην προάσπιση των γυναικών στον τομέα της ελευθερίας, ε, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης που είναι αυτό που αναζητούμε όλοι μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ καλή η συζήτηση που κάναμε για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Το χρονοδιάγραμμα ξεχάσαμε. Στις 5 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες. 5 Δεκάτου στις 12 το μεσημέρι. Ε, και προβλέπουμε να ψηφίσουμε στις 19 Οκτωβρίου στην Επιτροπή, στην έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Στρασβούργο. Και κατόπιν έχουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, στη 2η του Νοεμβρίου, στις 20, από τις 23 μέχρι τις 26. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Προχωράμε. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο 12. Έχουμε ένα προσκεκλημένο. Θα τον περιμένουμε λίγα λεπτά. Δεν έχει ακόμη προλάβει να φτάσει. Καλωσορίζω την κυρία Ντανιέλ Ρισάρ, προϊσταμένη στο τμήμα εκπόνησης πολιτικής. Με αυτό το policy department έχουμε ήδη καλή συνεργασία. Και η κυρία Ρισάρε θέλησε ήδη στην αρχή της θητείας να έρθει στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσει τις εργασίες τους. Είναι μια εξαιρετική αρχή για την ε, μελλοντική συνεργασία που θα έχουμε. Ε, είναι καλό το νωρίτερο δυνατόν να ενημερωνόμαστε Παρακαλούμε, κυρία Ντανιέλ Ρισάρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για αυτήν ε, ευγενική εισαγωγή. Συνήθως δεν εμφανίζονται οι υπηρεσίες εις ε, το Κοινοβούλιο αλλά στην προηγούμενη θητεία διαπιστώσαμε, ήμασταν μια νέα υπηρεσία ότι χρειάστηκε χρόνος για να αντιληφθούν οι προβλεφτές ε, πώς μπορούσαν να επωφεληθούν. Τα policy departments είναι υπηρεσίες έρευνας που προσφέρουν ε, ορισμένες υπηρεσίες στις κοινοβουλευτικές επιτροπές πέραν ε, του ό,τι κάνει η κυρία Μανιάνο και η ομάδα της ε, στη γραμματεία της ε, Επιτροπής. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα θέμα εσωτερικό ή εξωτερικό. Έχετε όλοι κάποιον προϋπολογισμό τον οποίο μπορούμε να δαπανίσουμε μόνο κατόπιν αποφάσεως του συντονιστών. Δεν μπορούμε δηλαδή να διασπαθήσουμε το δημόσιο χρήμα χωρίς να έχουν αποφασίσει οι συντονιστές. Οπότε ε, εάν πρόκειται για εξωτερικές αγορές γίνεται διαγωνισμός αλλά υπάρχουν δυνατότητες τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ε, θελήσαμε λοιπόν να σας δώσουμε ένα μέτρο με το οποίο θα μπορέσουμε ε, να χρησιμοποιήσουμε ονομαστικά και προσωποποιημένα τα γλωσσικά προφίλ των ευρωβουλευτών διότι θα πρέπει κάθε στοιχείο να προσφέρεται στην ε, μητρική γλώσσα το ενδιαφερομένου και για ό,τι δεν υπάρχει μεταφρασμένο λάβαμε υπόψη το δεύτερο, ε, τη δεύτερη γλώσσα τουλάχιστον. Ίσως φαίνεται λίγο πεπαλαιωμένο διότι αυτή τη στιγμή λαμβάνεται πολύ ωραία έγγραφα ή ε, ε, USB sticks αλλά το κλασέρ δεν χάνεται. Το έχετε και εμείς θα μπορούμε να προτείνουμε ενημερώσεις είτε διότι έχουμε επιπλέον πληροφορίες οι οποίες υιοθετήθηκαν ή θέλουμε να δώσουμε νέα τα οποία δεν υπήρχαν ε, προηγουμένως οπότε σας ε, στέλνουμε ένα μήνυμα στείλτε το τμήμα 1-1 και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Θα πρέπει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να μπορείτε να ε, αποφύγετε ότι δεν σας ενδιαφέρει, να τα πετάξετε. Με συγχωρείτε για το κινητό μου, πάντοτε χτυπάει στην κατάλληλη στιγμή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το κλασσάρ αυτό θα σας βοηθήσει, ότι θα είναι προσωποποιημένο, ότι δεν σας ενδιαφέρει μπορεί να πεταχτεί, θα κρατήσετε αυτά που σας ενδιαφέρουν προσωπικά. Εμείς ε, συγχρόνως συνεργαζόμαστε με τη γραμματεία, οπότε ένα θέμα που αναφέρεται στις ε, εργασίες ε, ερεύνης που αναφέρεται στην κυρία Μανιάνο θα σταλεί σε αυτήν, ό,τι αναφέρεται στην Επιτροπή θα σταλεί στη Σαβίνα. Θέλω να σας πω ότι αυτό το ίσως πεπαλαιωμένο στοιχείο ε, έχει μεταφραστεί και σε USB stick, δηλαδή αν δεν θέλετε να τρέχετε στο Στρασβούργο με το κλασέρ, μπορείτε να πάρετε το stick USB μαζί σας. Και τέλος ε, θέλω να παρουσιάσω την ε, ειδικό μας, την κυρία Κλέρ Ζαντά, η οποία επανέρχεται στην ε, Επιτροπή Γυναικών, διότι έγινε μία αναδιοργάνωση και η προηγούμενη υπεύθυνη πάει τώρα στις εσωτερικέ υποθέσεις και στη δικαιοσύνη και η Κλέρ είναι στη διάθεσή σας όταν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σε θέματα ερεύνης και με τα μεγάλη χαράς θα έχουμε τα σχόλιά σας διότι πρόκειται για μία δουλειά η οποία είναι πνευματικά σημαντική, υλικά πολύ ενδιαφέρουσα και ακόμη και αν έχετε αρνητικά σχόλια, προτιμώ να έχετε θετικά βέβαια, προσπαθήστε να αντιδράσετε γιατί η εμπειρία αυτή έχει ληφθεί από ένα τμήμα, δεν ξέρω αν θα γενικοποιηθεί, θα γενικευτεί, αλλά καλό θα ήταν να γενικευτεί αναλόγως με τις αντιδράσεις των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ελπίζω ότι δεν μακρηγόρησα τόσο όσο την προηγούμενη φορά. Σας ευχαριστούμε και για τις πληροφορίες και για το ιστορικό υπόβαθρο που εκθέσατε. Ευχαριστούμε για το υλικό που μας δώσατε. Φυσικά έχουμε πολλά πράγματα στη διάθεσή μας, ιστοσελίδες και τα λεπά. Αλλά αυτό το υλικό συνδέεται άμεσα με τις εργασίες μας και είναι πάρα πολύ πρακτικό, ξέρετε, να τα έχουμε όλα μέσα σε ένα ε, κλασέρ. Είναι όλα συγκεντρωμένα λοιπόν και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και το ίδιο θα νομίζω θα συμφωνήσουν μαζί μου και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ε, όταν θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτούς τους φακέλους που μας δώσατε. Υπάρχουν ερωτήσεις ήδη τώρα για το υλικό αυτό. Κυρία Κορνέλισον, ε, παρακαλώ. Um, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το τμήμα πολιτικών γιατί η πληροφορία αυτή και ο χάρτης είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα είναι χρήσιμο και το USB ε, ιδίως ε, για κάποιον σαν και μένα που είμαι καινούρια ξεκίνησα τον Ιούνιο διαβάζω τα πάντα και έτσι θα με βοηθήσει πολύ. Θα ήθελα να μας πείτε αν μπορείτε να μας ε, δώσετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα θέματα τα οποία επιλέγονται επί των οποίων εσείς προβαίνετε σε έρευνα διότι από ό,τι κατάλαβα η Επιτροπή αποφασίζει τα θέματα και μετά πρέπει να αποφασίσει ε, συγκεκριμένα πώς θα διατυπώσει τα ερωτήματα που θα τεθούν, τη μεθοδολογία ε, η οποία θα ακολουθηθεί για την έρευνα και θα ήθελα να ξέρω πώς όλα αυτά αποφασίζονται. Η κυρία Ρισάρ τώρα θα πάρει το λόγο για να μας απαντήσει. Ναι, βεβαίως, με τα χαράς. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω. Λοιπόν, να σας εξηγήσω πώς ε, γίνονται οι επιλογές. Οι επιλογές ε, των θεμάτων ε, φυσικά είναι θέμα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. σίγουρα τα μέλη της Επιτροπής θα μεριμνήσουν ώστε να γίνεται μια ορθή χρήση των ε, κονδυλίων. Είναι ζωτική σημασία στην πράξη να μην πληρώσουμε δεύτερη φορά μια μελέτη που ήδη έχει γίνει από κάποιον άλλον ε, για να βρούμε δεδομένα που είναι ούτως ή άλλως προσβάσιμα. Ο άλλος όρος είναι ότι δεν μπορεί μόνος του ή μόνη της μια βουλευτής να αποφασίσει να ζητήσει μια μελέτη. Πρέπει να υποβληθεί το αίτημα στους συντονιστές και να αποφασίσουν οι συντονιστές. Αν υπάρχει πληθώρα ε, αιτήσεων θα κληθεί να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες η Επιτροπή προς το παρόν. Ε, το πρόβλημα μας δεν ήταν τα κονδύλια, ήταν οι ανθρώπινοι πόροι. Η Κλέρ είναι μόνη της, το βλέπετε. Εγώ έρχομαι εδώ ως προϊστάμενη και έχω ε, πέντε επιτροπές και δεν θα με ξαναδείτε σύντομα. Η Κλέρ Ζαντά θα αναλάβει όλες τις μελέτες που χρειάζονται για την Επιτροπή των Γυναικών. Ε, ένα μέλος επιτροπής λοιπόν μπορεί να έρθει άμεσα σε επαφή μαζί μας αν θέλει να ζητήσει μια μελέτη ή να περάσει από τη Σαμπίνα. Μετά θα κάνουμε εμείς μια προκατακτική έρευνα αν ήδη έχει μελετηθεί το ζήτημα, πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Ορισμένες φορές, ε, παραδείγματος χάρη, στην προηγούμενη θητεία ε, μελετήσαμε ιδιαίτερο στο θέμα των γυναικών ΡΟΜ. Αλλά κάνοντας την προκατακτική αυτή έρευνα είδαμε ότι ήδη έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα για τις γυναίκες ΡΟΜ και ε, διαπιστώσαμε ότι οι έρευνες έφεραν ως επιτοπλίστων ε, επί της ε, οικονομικής κατάστασης ε, των γυναικών Ρώμων. Και αυτό που κάναμε ήταν να ομαδοποιήσουμε τα απορίσματα των διαφόρων ερευνών που είχαν γίνει. και ξαναλέω δεν είναι μόνο θέμα κονδύλιων, δεν ε, εντοπίζεται εκεί το πρόβλημα. Η ε, ανθρώπινη πόρη είναι μόνη της η Κλεζάντα, ε, δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες, δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της, οπότε εσείς θα αποφασίσετε ποιες είναι οι προτεραιότητες για την Επιτροπή και κάτι άλλο που δεν αντιλαμβάνονται εύκολα τα μέλη της Επιτροπής και μας κατηγορούν ότι είμαστε γραφειοκράτες, ενώ δεν είμαστε καθόλου, είναι ότι καθυστερούμε Μα ε, είναι, αυτό οφείλεται στο, στις ρυθμίσεις του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ε, ε στη σχετική νομοθεσία για τις ε, κρατικές συμβάσεις. Πρέπει πρώτα να γίνει η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, να γίνει όλος ο διαγωνισμός, να μεταφραστούν όλα σε όλες τις γλώσσες ε, μετά να γίνει μελέτη πρέπει και εμείς να αξιολογήσουμε τις μελέτες, να τις βαθμολογήσουμε. Ε, μετά πρέπει να πάρουμε την έγκριση για, την, ε, για τις δαπάνες. Παίρνουν χρόνο όλα αυτά, οπότε το λέω αυτό γιατί αν μας ζητήσετε κάτι για αύριο είναι απλώς αδύνατο να γίνει. Ε, ανάλογα με τη σημασία των ζητημάτων, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι για, τις, ε, για όλες τις μελέτες, συγκριτικές μελέτες ε, που καλύπτουν την Ένωση των 27 είναι χρονοβόρες και κοστίζουν πολλά χρήματα και απαιτούν πολύ χρόνο. Μόλις περατωθεί ε, η επαχθής ε, διαδικασία που συνεχίζει τώρα μέχρι το Δεκέμβριο, θα έχουμε έτοιμους τους εμπειρογνώμονες, θα τους στέλνουμε ένα δελτίο και θα τους ζητάμε τη συνεισφορά τους για ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο και η απάντηση θα μας έρχεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό για ένα συγκεκριμένο θέμα. Αλλά όταν είναι περίπλοκο το ζήτημα ή θέλουμε στοιχεία από τις 27 χώρες της Ένωσης, ε, δεν γίνεται να προσφύγουμε σε αυτήν την αναθεωρία θεωρημένη διαδικασία με τους εμπειρογνώμονες. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Η κυρία Κώστα ζήτησε το λόγο. Χαίρομαι που έχουμε αυτή την άμεση επαφή, διότι για μας είναι πολύτιμα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για το δώρο που μας κάνετε. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι εξής. Επειδή φαντάζομαι είναι πολύ σημαντική αυτή αυτός ο συντονισμός με την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής και τις μελέτες και καταλαβαίνω και το θέμα του χρόνου που απαιτείται. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον θα μπορούσαμε από τώρα να σκεφτούμε τουλάχιστον δύο θέματα που θεωρούμε ότι βρίσκονται ε, στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει η ένδια για του χρόνου, για παράδειγμα, και ο εθελοντισμός ε, για την μεθεπόμενη χρονιά. Ίσως λοιπόν από τώρα θα μπορούσαμε, τουλάχιστον και αυτά τα δύο πράγματα, ε, να σας τα εμπιστευτούμε αυτά, διότι οι γυναίκες και στους δύο τομείς αυτούς είναι μια πάρα πολύ ισχυρή πραγματικότητα και καλό θα ήταν να εμβαθύνουμε λίγο περαιτέρω σε αυτά. Επίσης, θεωρώ είναι και πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της συμφωνίας πλαίσιο, διότι επιτρέπει να έχουμε και ένα ε, σύνολο πυρογνωμένων και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, τι σχέση υπάρχει θετική, είναι παγιωμένη αυτή η σχέση με τα ερευνητικά κέντρα και τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Πού απευθύνεστε ε, και στην Ιταλία για παράδειγμα για να λάβετε πληροφορίες ε, τύπου ερευνητικά Ινστιτούτα, στατιστικά Ινστιτούτα ε, υπάρχουν ήδη σχέσεις σημαντικές με πυρογνώμενες και κρατημέλη ή μέσω των δικών σας ερευνητών ε, προχωράτε. Ευχαριστούμε κυρία Κώστα. Ε, κυρία Γησάχ, σας ξαναδίνω το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις της κυρίας ε, Κώστα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Μπορώ να απαντήσω λοιπόν σχετικά με την, τα κέντρα ερευνών. Διατηρούμε ως το δυνατόν περισσότερες επαφές με ως το δυνατόν περισσότερα κέντρα ερευνών με ορισμένους περιορισμούς. Πρώτον, είναι προφανές ότι όταν εργαζόμαστε σε επίπεδο ευρωπαϊκό δεν σημαίνει ότι την προτεραιότητα την έχουν τα κέντρα στις Βρυξέλλες αλλά ζητήσαμε τα κέντρα αυτά να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο δικτυωμένα διότι αν υπάρχει ένα δίκτυο στην Πούλια δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αλλά τώρα τα κέντρα ερευνών το ξέρουν και αναπτύσσουν διασυνδέσεις. Πώς θα επιλέγουμε βάσει της ε, ε, νομοθεσίας των δημοσίων αγορών. Μέχρι 60.000 ευρώ εντοπίζουμε ως το δυνατόν περισσότερα κέντρα που μπορεί να μας ενδιαφέρουν ε, σχετικά με την ποιότητα των, της δουλειάς τους και στέλνουμε μία μία πρόσκληση για να μας διατυπώσουν προτάσεις σε τουλάχιστον πέντε τέτοια Ινστιτούτα ερευνών. Πέντε είναι ελάχιστα, Αν έχουμε 25 ή αν εσείς έχετε να μας προτείνετε κάτι ενδιαφέρον, ευχαρίστως να μας το πείτε. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι θα επιλεγούν και έρχομαι τώρα στο δεύτερο μέρος. Άπαξ και επιλεγούν, δηλαδή μάλλον μετά από τις 60.000 ευρώ δεν επιλέγουμε κανέναν, είναι ανοιχτή επιλογή και πρέπει να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε περισσότερη διαφήμιση από την επίσημη εφημερίδα διότι τότε ε, όμως μας λέγουν ότι δίνουμε προνομιούχες προτάσεις και πληροφορίες σε ορισμένους ε, βέβαια κανείς ε, δεν κοιτάζει καθημερινά ε, την επίσημη εφημερίδα. Απάντω από 60.000 ευρώ πάντως σε δημόσιος διαγωνισμός. Και τα κριτήρια είναι κριτήρια επιλογής τα οποία αναφέρονται εις την προκήρυξη του διαγωνισμού υπάρχει κάποιος που κάνει τον αφελή έρχεται από κάποιο άλλο τομέα και μπορεί να κοιτάξει τα θέματα αντικειμενικά και ε, μετά ο υπεύθυνος ε, ε, επιτρέπει την δαπάνη, υπάρχει δηλαδή μία επιλογή ε, εσωτερική αλλά επιστημονική επαγρυπνούμε, ζητούμε από τους προβουλευτές ε, ε, να παρακολουθούν και να παρακολουθούν τη δημοσιονομική δαπάνη διότι αν εμείς δώσουμε μία πληροφορία σε λίγους προνομιούχους τότε εμείς θεωρούμαστε υπεύθυνοι Πρέπει λοιπόν να τους δείξουμε τις προδιαγραφές και εάν ε, το ε, στείλει σε κάποιον ο βοηθός ε, την πληροφόρηση πριν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα τότε ακυρώνεται ο διαγωνισμός μέχρι ότου να σταλούν οι φάκελοι καλώντας για να υποβάλουν προτάσεις δεν μπορεί να κυκλοφορήσει η πρόταση μελέτης. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένοι περιορισμοί που αναφέρονται στη διαχείριση των δημοσίων χρημάτων. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες και ευχαριστούμε και για το φάκελο με το υλικό που μας δώσατε. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία στο μέλλον. Προχωρούμε. Ανακοινώσει του Προέδρου. Έχω διάφορες σύντομε ανακοινώσεις. Κάναμε συνεδρία των συντονιστών σήμερα το πρωί. Αρχίσαμε σε 9 και λάβαμε τις αποφάσεις εκεί. Αποφασίσαμε να κάνουμε μία έκθεση για το ρόλο των γυναικών στη γυράσκουσα κοινωνία. Ανατέθηκε στο ΕΛΚ αυτή η έκθεση. Επίσης, σε μία γνωμοδότηση θα εκδώσουμε για τα μέτρα καταπολέμησης του καρκίνου. Οι σοσιαλιστές ανέλαβαν αυτή τη γνωμοδότηση. Επίσης, αποφασίσαμε ε, για τα πλήρη και για τα αναπληρωματικά μέλη για το Φόρουμ των Εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Δύο Φύλων. Η απόφαση έχει ως εξής. Πλήρη μέλη θα είναι η κυρία Λίζ Κέλλη και η κυρία Βίλε Μερόιγκροκ. Διορίστηκαν ως πλήρη μέλη, λοιπόν, οι κυρίες αυτές. Αναπληρωματικά μέλη είναι η κυρία Μανταριάγκα Μπαστούρη και η κυρία Λίζη Γκρένερ. Αυτή ήταν η έκβαση της ψηφοφορίας των συντονιστών σήμερα το πρωί. Επίσης, απο, πήραμε αποφάσεις για τις ακροάσεις που θα γίνουν ε, στα πλαίσια του προγράμματος εργασιών της Επιτροπής. Θα διοργανωθούν οι εξή ακροάσεις λοιπόν. Η πρώτη είναι προς μία νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων. Θα είναι μία από τις ε, σημαντικότερες εκδηλώσεις της Επιτροπής μας στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος εργασιών. Αυτή η νέα στρατηγική λοιπόν και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να αποφασίσουμε διάφορα συγκεκριμένα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στη στρατηγική αυτή. Θα αποτελέσει επίσης αυτή η ακρόση μια πλατφόρμα για τις μελλοντικές εργασίες ε, της Επιτροπής μας στον τομέα αυτό. Δεύτερη ακρόαση Το 2010 είναι το έτος καταπολέμησης της ένδυας ε, και του κοινωνικού αποκλεισμού και λόγω τους ευρεία συνένες επιλέχθηκε αυτό ως θέμα για τη δεύτερη ακρόαση. Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό το ζήτημα. Η τρίτη ακρόαση για την οποία συμφωνήσαμε είναι για την κοινωνική ένταξη των γυναικών που ανήκουν σε, εθνοτικές, σε εθνικές μειονότητες. Αυτές τις τρεις αποφάσεις πήραμε για τις ακροάσεις. Επιπροσθέτως, συζητήσαμε ποιο θα είναι το θέμα για την Διεθνή ημέρα γυναικών Ε, ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε για να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε και τις εργασίες μας και αποφασίσαμε λοιπόν ότι το θέμα θα είναι η βία κατά των γυναικών και έχουμε ήδη αποφασίσει πότε θα εορταστεί η Διεθνής ε, ημέρα γυναικών και επιλέχθηκε αυτό το θέμα ε, της βίας κατά των γυναικών διότι η επόμενη Προεδρία, η Ισπανική Προεδρία το πρώτο εξάμεινο το 2010 ε, ε, έχει ορίσει αυτό το θέμα της βίας κατά των γυναικών ως προτεραιότητα ήδη στο πρόγραμμά της. Αποφασίσαμε επίσης ε, ποια ταξίδια θα γίνουν από τις αντιπροσωπείς επιτροπής μας για το 2010. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που θα σας δώσω από την σημερινή συνεδρία των συντονιστών. Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη διάσκεψη του ΟΗΕ που θα γίνει σε αρχές Μαρτίου για την ε, συνέχεια που δίνεται στην ε, διάσκεψη του Πεκίνου, δηλαδή Πεκίνο συν 15. Συμφώνησαν οι συνάδελφοι ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε και στη διάσκεψη του ΟΗΕ. Αποφασίσαμε επίσης ε, να πάει μια αντιπροσωπεία στη Βουδαπέστη λόγω της μελλοντικής Ουγγρικής Προεδρίας. Είχαμε αποφασίσει ότι θέλουμε να γίνουν αυτές οι επισκέψεις για να προετοιμάσουμε την επιχείμενη ε, Ουγγρική Προεδρία. Επίσης, ε, στο Ινστιτούτο Ισότητας των Δύο Φύλων, Gender Institute, ε, θα ε, πάει μία αντιπροσωπεία τον Μάιο-Ιούνιο του 2010. Ελπίζουμε κάθε δύο χρόνια να έχουμε τη δυνατότητα να επισκεπτόμαστε αυτό το Ινστιτούτο λόγω του κοινού συμφέροντος που έχουμε. Είναι προς συμφέρον αμφωτέρων των πλευρών να έχουμε στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο. Επίσης, Ισλανδία, άλλη μια αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Ισλανδία. Είναι επίκαιρο το θέμα, διότι Όπως μας είπαν οι συντονιστές σήμερα το πρωί θεωρούν ότι είναι ε, καλή πρόταση για ε, ε ταξίδια του προσωπίας η Ισλανδία λόγω της ε, αίτησης προσχώρησης. Ε, φυσικά, ε, για όλες αυτές τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους συντονιστές θα πάρετε και θα σας μοιράσουμε και τα πρακτικά. Υπάρχει κάτι υπό τα διάφορα, περνώ δηλαδή στο σημείο 14. Εάν όχι, 15. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 19 Οκτωβρίου θα συνεδριάσουμε στο Στρασβούργο. Είναι μια έκτακτη συνεδρίαση όπου θα γίνει ψηφοφορία και όπου θα συναντηθούμε με την Επίτροπο Βάλινστρομ στις 19 Οκτωβρίου. Και ε, στις 4 Νοεμβρίου θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες. Ε, θα περάσει πολύ καιρός μέχρι την επόμενη συνεδρίαση Επιτροπής μας ε, στις Βρυξέλλες from the policy department. They can leave it here and we will have it sent. και κάτι άλλο. Ε, για τα μέλη που δεν ε, μπορούν να πάρουν μαζί τους το φάκελο του Policy Department, να το αφήσετε παρακαλούμε πάνω στο τραπέζι. Κάποιος ε, θα μεριμνήσει για να σας το δώσουμε στο γραφείο σας. Στο φέρουμε στο γραφείο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειές σας και χθες και σήμερα για να γίνεται με επικοδημητικό τρόπο η συζήτηση. Ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερως για τη συνεργασία με όλα τα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τη γραμματεία της Επιτροπής γιατί είχε προετοιμάσει με εξαιρετικό τρόπο τη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος ευγενικά ευχαριστεί και τους Ερμηνείς.